Είναι, υπάρχει ελληνική μετάφραση, υπάρχει. Λοιπόν, καλημέρα σας. Είμαστε έτοιμοι. Μια μικρή αλλαγή στην σειρά των δύο πρώτων θεμάτων. Δεν υπάρχουν, νομίζω, ανακοινώσει από τη μεριά της, του, του Προεδρείου. Όταν θα έρθει η κυρία... η πρόεδρος θα μιλήσουμε γι' αυτό. Θα ξεκινήσουμε με το 13 που αφορά στην έκθεση για, την ετήσια, για τον Ευρωπαίο Μεσολαβητή. Η κυρία Γιώτοβα το ζήτησε και παρακαλώ να ε, μας εκθέσει τις απόψεις της για την έκθεση του 2010. Ευχαριστώ. Благодаря, госпожо председател. Годишният доклад за дейността на омбудсмана показва... Η ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή δείχνει τον εξαιρετικό επαγγελματισμό όλης της ομάδας του κυρίου Διαμαντούρου. Οι υποθέσεις έχουν να κάνουν με θέματα διοικητικά και προσπαθεί η υπηρεσία αυτή να προστατεύσει τους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό το άτομο που κατέχει τη θέση αυτή να γνωρίζει τους θεσμούς και τη λειτουργία τους. Θα ήθελα πραγματικά λοιπόν να συγχαρώ όλη την ομάδα, του συνεργάτες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την στρατηγική και τις κατευθύνσεις που ακολούθησαν καθ' όλη τη διάρκεια της εντολής τους. Σήμερα ο στόχος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι με ανοιχτό τρόπο, με διαφανή τρόπο να επιτευχθούν οι διοικητικές διαδικασίες. Διαδικασίες οι οποίες θα είναι εύκολες όσον αφορά την πρόσβασή τους για τους Ευρωπαίους πολίτες. Βασιζόμαστε πάντα στην, στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το 2010 ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής συνέχισε να ασκεί ε, την εξουσία του με ένα εξαιρετικά ισορροπημένο τρόπο. Έδειξε ότι πραγματικά πάνω απ' όλα βρίσκονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Έδειξε επίσης ότι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εργάζονται προς συμφέρον των πολιτών. 333 ε, έρευνες έγιναν το 2010. Δημιουργήθηκε και μία ιστοσελίδα διαδραστική η οποία, στην οποία καταχωρούνται οι αναφορές. του ε, το 2009 υπήρξαν 3.900 ε, αναφορές. Το 2010 ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 3.600. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι είχαν αδυναμίες οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και δεν μπόρεσαν να καταχωρήσουν περισσότερες ε, αναφορές. Αντίθετα, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή αυτή η εξαιρετική πρωτοβουλία, αυτή η διαδραστική σελίδα επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να ενημερώνονται με σωστό τρόπο όσον αφορά τις αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν τα μέσα που διαθέτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ και πολλές ε, συνεδριάσεις η συζήτηση που έγινε εδώ αφορά τις αρμοδιότητες και τον τρόπο που λειτουργεί ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Και βεβαίως χρειάζονται περισσότερα μέσα για την περαιτέρω ανάπτυξη της, ε, του ιστοτόπου. Γιορτάζουμε σήμερα την 15η επέτειο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών έχει αυξηθεί χάρη στην ανεξαρτησία αυτού του θεσμού, χάρη στο δημοκρατικό έλεγχο που ασκείται από μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά τα 15 χρόνια λειτουργίας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή του έδωσαν τη δυνατότητα να υλοποιήσει ποιες είναι να υλοποιήσει πολύ σημαντικά επιτεύγματα, να διαπιστώσει ποιες είναι οι αδυναμίες λειτουργίας των θεσμών καθώς και οι αδυναμίες που υπάρχουν στη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Παρόλα αυτά, ο αριθμός των ε, αναφορών όσον αφορά παραδείγματο χάρη την ε, πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι εξαιρετικά υψηλός. Η πρόσβαση στις πληροφορίες πολλές φορές δεν είναι εφικτή. Ακόμα και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχουν πρόσβαση. Άρα δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια στις ε, διεργασίες και στα έγγραφα του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρουσία εκπροσώπων του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου, οι Ευρωβουλευτές, θα πρέπει λοιπόν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που παραδείγματο χάρη χρησιμοποιούν, επικαλούνται οι συνεργάτες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για να ε, απορρίψουν μία αναφορά δίνονται απαντήσεις ε, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό αποτελεί ένα ξεχωριστό τμήμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Διαμαντούρο καθότι πάντα έδειξε προθυμία συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντα για το καλό των Ευρωπαίων πολιτών. Θεωρώ ότι αυτές οι επικοδημητικές σχέσεις θα πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα για όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ε, ευχαριστώ πολύ την κυρία Γιώτοβα. Ε, η κυρία Άουκεν ζήτησε να μιλήσει πριν από την Επιτροπή γιατί έχει μια άλλη συμμετοχή κάπου αλλού. Παρακαλώ κυρία Άουκεν. Ja, tusind tak, fru formand, øh, og tusind tak, fordi jeg fik lov til at få ordet først. Jeg skal hen til den konference, hvor også vores formand er til stede. Ευχαριστώ που δίνετε το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ για αυτή την ε, εξαιρετική έκθεση. Μιλήσατε για διαφάνεια. Είναι εξαιρετικό. Ως κείμενο, το Κοινοβούλιο θα πρέπει τώρα να προσεγγίσει ώστε να το περισσότερο τους πολίτες για να κατανοήσουν τον το δικό μας ρόλο, το ρόλο του Κοινοβουλίου ως διαμεσολαβητή. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να απογραμμίσουμε. Αυτό που αποκαλούμε good administration, μια καλή διαχείριση, η ορθή διαχείριση, είναι ουσιώδες στοιχείο της ε, λειτουργίας μας. Στο μέτρο του δυνατού, ε, μια κοινή διαχείριση, θα είμαι σύντομη, θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 2098 του, ε, της συνθήκης της, ε, της θα αναφερθώ σε αυτό το άρθρο στα αγγλικά για να τονίσω αυτό που είναι σημαντικό στην ε, έκθεσή μας. Το λέω στα αγγλικά. θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη ενός μια ανοιχτής, ε, επαρκούς και ε, ανεξάρτητης ευρωπαϊκής ε, διαχείρισης. Σύμφωνα με τα, τις διατάξεις του άρθρου 336, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με τον κανονισμό και με την νομοθετική διαδικασία, θα καθιερώσει διατάξεις προς αυτό το σκοπό. Αυτό θέλω να τονιστεί ακόμα περαιτέρω στην ε, έκθεσή σας. Έτσι θα είναι μια πραγματικά πάρα πολύ καλή έκθεση και έτσι να σας ευχαριστήσω από αυτή την ευκαιρία ε, και τον Ευρωπαϊκό Μεσολαβητή για το έργο του. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Εμεί ευχαριστούμε κυρία ε, Άουκεν. από την Επιτροπή η κυρία Κώστα Ρώσα. Παρακαλώ. Ε, je passe d'abord la... Καταρχήν θα δώσω το λόγο στον επικεφαλής της υπηρεσίας για τη διαφάνεια και την πρόσβαση στα έγγραφα, ο οποίος πρέπει να φύγει, όπως και η κυρία Όκεν, γιατί έχει μια άλλη συνάντηση στις 10. Και κατόπιν θα πάρω εγώ το λόγο και θα κάνω κάποια γενικότερα σχόλια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, που μου δίνετε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Γιώτοβα για την ε, εργασία της που περιέχει σημαντικό αριθμό παρατηρήσεων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Επιτροπή. Εκφράζετε την άποψή σας και πιστεύω ότι οι συνάδελφοι ε, μετά από μένα θα κάνουν κάποια επιπλέον σχόλια. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα που αφορά τη διαφάνεια καθώς και την πρόσβαση στα έγγραφα. Εδώ υπάρχουν ε, δύο ή τρεις παρατηρήσεις οι οποίες ε, χρήσουν απάντησης οι σχέσεις μας με τον διαμεσολαβητή είναι πολύ καλές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει η ειλικρινή αυτή συνεργασία να αναπτυχθεί περαιτέρω με τον διαμεσολαβητή. Η ειδική έκθεση την οποία αναφέρετε και για την οποία κάνετε κάποια σχόλια οδήγησε σε μια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Δεν θα επανέλθω λοιπόν στις λεπτομέρειες αυτή τη ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα απλώς να πω ότι καταρχήν η Επιτροπή αναγνωρίζει στην συγκεκριμένη αυτή περίπτωση ότι όντως υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι οι καθυστερήσεις αυτές σημαίνουν ότι αγνοούμε τις ε, αρμοδιότητες του διαμεσολαβητή. Εξηγήσαμε αυτή την καθυστέρηση η οποία οφείλεται στην ε, βούληση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που διαθέτει έτσι ώστε να ε, δημοσιευθούν όλα τα στοιχεία αυτά. Και αυτό μας οδηγεί σε μια γενικότερη παρατήρηση όσον αφορά τη διαφάνεια και την πρόσβαση στα έγγραφα. Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση, σαν και αυτή που συζητούμε σήμερα, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τον απόϊχο τα σχόλια, της παρατηρήσεις που ακολουθούν μια τέτοια υπόθεση, οι οποίες όμως ουσιαστικά κρύβουν την μεγάλη εμβέλεια των απαντήσεων που δίνει διαρκώς καθημερινά, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα η Επιτροπή όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να υπογραμμίσουμε ότι πάνω από το 80% των ε, αιτήσεων για πρόσβαση σε έγγραφα ικανοποιούνται ήδη από την πρώτη αίτηση. Και με την ε, διαδικασία της ε, δεύτερης δυνατότητας αίτησης, όλες οι αρνητικές απαντήσεις σε μεγάλο βαθμό ικανοποιούνται. Και πολύ σύντομα θα έχετε και τα στατιστικά στοιχεία για το 2010. Θα δείτε λοιπόν ότι όντως στη δεύτερη αίτηση, στην έφεση αν θέλετε, μετά από μια πρώτη αρνητική απάντηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ικανοποιεί τα αιτήματα. Είμαστε λοιπόν περήφανοι όσον αφορά την πολιτική μας σε θέματα διαφάνειας στην Επιτροπή. Πολλοί λένε ότι είμαστε πραγματικά σε εξαιρετικά καλή σειρά όσον αφορά την πολιτική μας σε θέματα διαφάνειας. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πούμε. Όπως ε, την ίδια ώρα αναγνωρίζουμε κάποιες ε, αδυναμίες ή κάποια σφάλματα που όλες οι διοικητικές υπηρεσίες γνωρίζουν στην καθημερινή τους λειτουργία. Αυτή λοιπόν η ειδική έκθεση είναι εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας και αυτό πρέπει να πούμε στους Ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει να είμαστε σε θέση να πούμε ότι όταν διαμαρτύρονται οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες, αν κοιτάξουμε καλά τις περιπτώσεις οι οποίες τελικά φτάνουν μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τις περισσότερες περιπτώσεις λοιπόν διαπιστώνουμε ότι δεν πρόκειται για πολίτες. Πρόκειται για δικηγορικά γραφεία τα οποία τροφοδοτούν φακέλους και υποθέσεις για να φτάσουν μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μα αυτό είναι θεμητό. Είναι κάτι που το επιτρέπει το κοινοτικό δίκαιο. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι όταν αναφέρουμε τις υποθέσεις αυτές και τα στατιστικά στοιχεία για να ξέρουμε ε, για τι θέματα μιλάμε. Αυτά ήθελα να πω κυρία Πρόεδρε για την ειδική αυτή έκθεση. Επίσης, όσον αφορά την νομοθετική διαδικασία που αφορά την πρότασή μας για αναθεώρηση του κανονισμού, η οποία έχει υποβληθεί από το 2008. Το 2008. Η πρόταση αυτή για αναθεώρηση του κανονισμού έχει υποβληθεί στο Κοινοβουλίο και στο Συμβούλιο και η Επιτροπή έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή υπέβαλε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ένα σύνολο προτάσεων για να ενσωματωθεί η νομολογία, για να λάβουμε υπόψη μας την μέχρι τώρα εμπειρία και για να προσαρμόσουμε τη συνθήκη, τον κανονισμό μάλλον στη συνθήκη. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, έχουμε συμμετάσχει σε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις για τον κανονισμό αυτό δεν μπορούμε όμως να ξαναπάρουμε το λόγο αυτή τη στιγμή, καθότι δεν γνωρίζουμε, η Επιτροπή δεν γνωρίζει ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάποια πράγματα ακούστηκαν. Υπάρχουν 90 τροπολογίες. Υπάρχει ένα κείμενο που προετοιμάζεται από μέρους του Κοινοβουλίου. Αυτό όμως δεν είναι η επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν δεν μπορεί να υιοθετήσει μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου καινούρια από τη στιγμή που δεν γνωρίζει ποιο είναι το περιβάλλον. Αυτό είπα λοιπόν και χτες και σε μια άλλη επιτροπή και πραγματικά ο κανονισμός 1049 στον οποίο μπορούν να προσθεθούν πάρα πολλά στοιχεία το θέμα αυτό μπορεί να γίνει πολύ πιο περίπλοκο. Ο κανονισμός 1049 μπορεί να εμπλουτιστεί με θέματα που αφορούν τη διαφάνεια, με άλλες διαδικασίες, όπως η ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παραδείγματο χάρη. Όταν μιλούμε για την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα θέμα το οποίο είναι θεμητό, το οποίο απαιτεί περισσότερη επεξεργασία, εδώ ξεπερνάμε το κανονισμό 1049 που αφορά την δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες και στα έγγραφα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί. Στις 28 Ιουνίου θα υπάρξει μία συνάντηση μεταξύ του Αντιπροέδρου Σέλκοβιτς και του εισηγητή επί της ουσίας, αλλά και όλους τους άλλους εισηγητές που έχουν αναλάβει τις γνωμοδοτήσεις, έτσι ώστε να αποσαφινιστεί λίγο το θέμα. Ελπίζω ότι η συζήτηση αυτή θα είναι επικοδομητική με σκοπό να αυξηθεί η διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελε κάποιος από τους συναδέλφους να μιλήσει για το θέμα. Ε, Καρό καταρχήν για την πρωτοβουλία να συζητήσουμε για θέματα που αφορούν στη διαφάνεια στο νομοθετικό, στην νομοθετική της διάσταση και δύο παρατηρήσεις ε, και στις δύο περιπτώσεις τις οποίες αναφερθήκατε και στην ειδική έκθεση της κυρίας Γιώτοβα και στην, ε, έκθεση για το 2010 των πεπραγμένων και στην ειδική έκθεση περιέργως έχω εμπλακεί ε, χαίρομαι ότι αναγνωρίζετε πως ήταν μια ειδική περίπτωση η καθυστέρηση η περίεργη αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα επίσης ότι το αποτέλεσμα της ειδικής αναφοράς του διαμεσολαβητή ε, ενεργοποίησε λίγο περισσότερο ε, ε, το τμήμα προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί απέναντι σε αυτό που λέμε διαφάνεια και πρόσβαση στα έγγραφα από τη μεριά των πολιτών. Επομένως θεωρώ ότι συνέβαλε μάλλον η ειδική έκθεση του διαμεσολαβητή και προς αυτή την κατεύθυνση της καλύτερης συνεργασίας ανάμεσα στους δύο θεσμούς. Και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι η κυρία Γιώτοβα ε, ε, επενεί τον θεσμό και τη δράση του διαμεσολαβητή ειδικότερα και της ομάδας του ε, ότι στην ουσία επεκτείνει τον έπαινο και την αποτελεσματικότητα που είχαμε διαγνώσει και στην προηγούμενη έκθεση για το 2009 που ήταν ομολογουμένως η πρώτη μου επαφή με το Ευρωκοινοβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τη δουλειά του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή απέναντι σε οποιασδήποτε δυσκολίες με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος και ευχαριστώ πολύ την κυρία Γιώτοβα για, ε, την έκθεση με την οποία συνέταξε. Euh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από την πολύ σημαντική αυτή παρέμβαση την σημαντικότερη θα έλεγα που αφορά το θέμα αυτό. Ο συνάδελφος είναι ειδικό για θέματα διαφάνειας. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Πρόκειται για μια εξαιρετική έκθεση που αφορά την ετήσια έκθεση του διαμεσολαβητή. Είναι πολύ ευανάγνωστη και η δομή αυτής της έκθεσης ήδη ήταν αντικείμενο σχολείων από μέρους της Επιτροπής πριν από ένα μήνα. Θέλουμε για άλλη μια φορά να επαναλάβουμε να υπογραμμίσουμε την πολύ στενή συνεργασία που έχουμε με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και με τους συνεργάτες του. Στην έκθεση του Διαμεσολαβητή υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που αφορά τις επαφές μεταξύ της ομάδας του και των υπηρεσιών της Επιτροπής. Είμαστε λοιπόν σε συνεχή και μόνιμο διάλογο. 375 απαντήσεις ε, δόθηκαν από μέρους της Επιτροπής των διαμεσολαβητή. περίπου 40 απαντήσεις το μήνα, αν δεν μετρήσουμε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό, αν θέλετε, ε, ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Αυξήθηκαν οι προσφυγές, οι μνήσεις προς την Επιτροπή. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η αντιμετώπιση από μέρους της Επιτροπής ήταν χειρότερη πέρσι. Απλώς όπως αναφέρει και η συγγήτρια, η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω του ιστοτόπου βοήθησε τους Ευρωπαίους πολίτες να μην συγχέουν τις αρμοδιότητες του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή και κάποιων άλλων ευρωπαϊκών θεσμών ε, στους οποίους μπορούν επίσης να αποτανθούν για να επιληθούν κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Υπάρχουν και κάποιες άλλες βεβαίως παρατηρήσεις πολύ αυστηρές θα έλεγα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές όμως μειώνονται και αυτό μας δείχνει ότι χάρη στη δράση του διαμεσολαβητή και στην συνεργασία της Επιτροπής η κακή διαχείριση μειώνεται. Βελτιώνεται η λειτουργία των υπηρεσιών μας και αυτό είναι μια καθημερινή, αν θέλετε, προσπάθεια εκ μέρους μας, μια καθημερινή προσπάθεια των διευθυντών, των συνεργατών τους. Καθημερινά κοιτάμε τι δυνατότητες υπάρχουν για επίλυση των υποθέσεων αυτών χωρίς να φτάσουμε στο δικαστήριο Η ιδιαίτερα για περιπτώσεις που δίνουμε έναν φάκελο, μια υπόθεση σε κάποιον ο οποίος είναι εντελώς εκτός αυτής της υπόθεσης για να μπορέσει με αμερόληπτο τρόπο να δώσει την άποψή του. Βεβαίως ξέρετε ότι το προσωπικό δεν είναι αρκετό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν μπορούμε να αυξήσουμε το προσωπικό μας. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε με το υπάρχον προσωπικό. Με μεγάλη χαρά είδαμε την κυρία Γιώτοβα η οποία αναφέρθηκε στην 15η επέτειο του θεσμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Συγχαίρουμε και εμείς τον κύριο Διαμαντούρο. Η νέα στρατηγική που υιοθέτησε είναι εξαιρετικά σημαντική και πιστεύουμε ότι η μελλοντική δράση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, η κατανόηση και η συνεργασία με τους άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η νέα στρατηγική, η νέα διαφάνεια, σίγουρα θα μας οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στις δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά την έννοια της ε, δημόσιας υπηρεσίας. Παρόλο που υπάρχει βεβαίως ο κώδικας συμπεριφοράς και το θέμα του κανονισμού, τα οποία βεβαίως θα πρέπει να επεξεργαστούμε περαιτέρω. ο διαμεσολαβητής και η εισηγήτρια δεν αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω και τον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή και την εισηγήτρια για την εξαιρετική τους εργασία. Ελπίζω η συνεργασία μας να είναι εξίσου καλή και ίσως και καλύτερη στο μέλλον. Πολύ απλώς να χαίρομαι ότι ενισχύεται ο θεσμός του Διαμεσολαβητή και προς τη μεριά της ε, Επιτροπής όσο περνάει ο καιρό και αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην, ε, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς γενικότερα. Ε, ευχαριστώ λοιπόν και την εισηγήτρια και, τα, τους εκπροσώπους από την Επιτροπή. Γυρνάμε πίσω στο θέμα 12 που αφορά στις κατευθυντήριες γραμμές ε, του προϋπολογισμού για το 2012 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο ε, ο κυρία Κόχ Μέρλιν δεν θα μπορεί να συμμετάσχει λόγω ασθενείας σήμερα. Ο κύριος Γιάρ ε, ανέλαβε να παρουσιάσει την εισήγηση για την γνωμοδότηση. Äh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να προσθέσω κάτι για το προηγούμενο θέμα, γιατί σήκωσα το χέρι και δεν με είδατε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια η συνεργασία με το διαμεσολαβητή είναι αξιέπαινη. Έχουμε σφυριλατήσει καλή συνεργασία. Εγώ είμαι ανάμεσα σε εκείνους που τα παράπονα του πολίτη για διοικητικά θέματα τα βλέπει ως θετικό δείγμα. Θα ήταν χειρότερο να μην είχαμε κανένα παράπονο. Η διοίκηση εξυπηρετεί τον πολίτη και όχι αντίστροφα και χρειάζεται feedback, ανάδραση, διάλογος με τον πολίτη που θα μας ενημερώσει αν κάτι δεν λειτουργεί καλά. Η αδιαφορία θα ήταν χειρότερη. Θεωρώ θετικό τον διάλογο με τον πολίτη, ο οποίος πολλές φορές δικαίως, άλλες φορές αδίκως παραπονείται για πράγματα που επιδέχονται βελτιώσεων. Δεύτερον, για τη διαφάνεια και την προστασία των δεδομένων. Περίπλοκο θέμα πρέπει να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι και εδώ είμαστε σε δρόμο καλό γιατί θα βρούμε μια διαδικασία που θα είναι δίκαιη και για τα δύο μέρη. Η διαφάνεια είναι καλό πράγμα, αλλά και απ' την άλλη θα πρέπει να προσέχουμε και την προστασία των δεδομένων. Δεν μπορούμε να την απορρίψουμε. Τρίτη παρατήρηση. Η Κομισιόν σωστά είπε ότι στο άρθρο 1049 ε, συμφωνεί με το, την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι και εμείς, αυτή, αυτή είναι μια αναφορά δηλαδή, ε, ότι πρέπει να εργαζόμεθα και να παίρνουμε αποφάσεις. Επίσης, βαστα, η, για την πρόταση της κυρίας Κοχμέριν τώρα, η κυρία Κοχμέριν δυστυχώς ασθενεί και με παρακάλεσε ο Σκιώδης να παρουσιάσω την έκθεση. Ευχαρίστως δέχτηκα γιατί γενικά μπορούμε να πούμε ότι στην ομάδα οι συγητές και οι Σκιώδης δεν εντόπισαν μεγάλα προβλήματα. Υπάρχει υψηλού βαθμού συνένεση για τα βασικά τώρα χαρακτηριστικά του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2012 μέτρια αύξηση του συνόλου 47% αύξηση κατά 0,47 σε 9 δίστε 400 κάτι εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ε, λαμβάνει υπόψη και τη δημοσιονομική πειθαρχία γιατί πέρσι ήταν πολύ ψηλότερες οι αυξήσεις. Στο πολιετές δημοσιονομικό σχέδιο συμπεριελήφθη συστηματική αναθεώρηση όλων των γραμμών του προϋπολογισμού για λόγους δημοσιονομικής αποτελεσματικότητας τα προγράμματα και τα έργα που μας ενδιαφέρουν μπορεί να σχεδιάζονται σε πολυετή βάση και μπορούμε εδώ να έχουμε σε 16 μέχρι 32 γραμμές του προϋπολογισμού εξοικονομήσεις. Τέλος, ε, ε, συμπεράσματα Προτείνομαι να ε, να εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού ως έχει η Επιτροπή. Επίσης ο διαμεσολαβητής μας υπέβαλε μια δημοσιονομική πρόταση η οποία λαμβάνει υπόψη τη σημερινή οικονομική κατάσταση και δεν προβλέπει σημαντικές δημοσιονομικές αυξήσεις. Καλό πράγμα είναι αυτό. Τρίτον, ο διαμεσολαβητής είναι σημαντικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου περί της αποδοχής της ίδιας της Ένωσης από τους πολίτες και ο θεσμός αυτός θα πρέπει να ενισχυθεί και με να πρικοδοτηθεί με κατάλληλους πόρους. Τέταρτον, χαίρομαι που θα έχουμε την ανταλλαγή απόψεων μαζί σας και με τους ε, σκιώδεις και βεβαίως είμαι ανοιχτό σε επικοδομητικές προτάσεις. Αυτά είχα να σας πω εξ ονόματος και της κυρίας Κοχμέριν. Ε, παρακαλώ κύριε Γιάννα να τα μεταφέρετε. Ε, θέλει κάποιος συνάδελφος. Α, η κυρία Κώστα Ρόζα από την Επιτροπή. Όχι, δεν έχω κάτι να προσθέσω από αυτού. Ευχαριστώ. Να ενημερώσω ότι για τις ε, τροπολογίες ε, τέρμινους είναι το 23, 23 Ιουνίου μέχρι τις 6 το απόγευμα και ε, για την προηγούμενη αναφορά για τη κυρία Γιώτοβα πάει στις 24 Ιουνίου μέχρι, μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έχουμε μια μικρή αναστάτωση ε, μετακίνηση θεμάτων. Επειδή η κυρία Ματσόνη θα ήθελε να είναι στο, ε, στη συζήτηση του υπαριθμών 14 ε, προχωρούμε στην ε, υπόθεση στην περίπτωση αριθμός 15 ε, η αναφέρουσα είναι παρούσα παρακαλώ λοιπόν, αφορά την αναφορά του κυρίου Σαλβαντόρ Λόπες Φλωρένσιο, Ισπανικής Ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης Χονδρεμπόρων Ιχθείων Ελμπαράνκο, σχετικά με το μονοπόλιο της Μερκασεβίλα στο χονδρεμπόριο Ιχθείων. παρακαλώ την ε, προσώπηση, την κυρία την αναφέρουσα. Α, είναι ο κύριος. Ο κύριος, ο Φορέντζη. Ο κύριος παρακαλώ. Sí. Sí, Ευχαριστώ. Καλημέρα. Αρχικά θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ και 25 χρόνια. Είμαστε ήχθιεύοροι στην κεντρική αγορά της Σεβίλης. Το Δημαρχείο Μα υποχρεώνει ε, να αποδεχθούμε ορισμένες υποχρεώσει και αν δεν τις αποδεχθούμε ε, θα χάσουμε την άδειά μας. Έτσι ε, υποχρεώμαστε, υποχρεώμαστε να καταβάλουμε 3,6% των ημερήσεων αποδοχών μας και αυτό μας επιβάλλεται από το Δημαρχείο και δεν είναι μοναδική η δική μας περίπτωση. Αυτό ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά αφορά μόνο τη δική μας αγορά, όχι στις υπόλοιπες, ας πούμε στην κρεταγορά ή σε άλλες αγορές. Ε, αυτό έχει τις εξής ε, επιπτώσεις. Μας αποτρέπει από το να μεταφέρουμε τα ε, εμπορεύματά μας στην περιοχή πώλησης. Δεν μπορούμε να εκδίδουμε τιμολόγια και έτσι παραβιάζουμε το, το κοινοτικό δίκαιο. Η Μερκασεβίγια είναι αυτή που εκδίδει τα τιμολόγια και έτσι έχει πρόσβαση και σε όλα τα ευαίσθητα ε, δεδομένα που αφορούν τις επιχειρήσεις μας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποδεχόμαστε επιταγές ή καθυστερημένες πληρωμές κτλ. Ε, υπάρχει λοιπόν μια προμήθεια 0,10% και δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τους ε, ε, υπαλλήλους της Μαρκασεβίγια. Υποχρεούμαστε να έχουμε εκείνου δηλαδή, οι οποίοι δεν είναι καν υποχρεωμένοι να είναι φιλικοί απέναντι στους πελάτες μας. Επίσης δεν έχουμε την δυνατότητα να συνάπτουμε συμβάσεις με τους ε, εργαζομένους μας. Έχουμε λοιπόν τον Ισπανό διαμεσολαβητή, ο οποίο ε, ε, εξέδωσε μια απόφαση για αυτό το ζήτημα πριν από μερικά χρόνια, είπε ότι υπήρχε ε, παραβίαση των δικαιωμάτων μας αλλά και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Η μερικασεβίγια λοιπόν και το ε, Δημαρχείο παραβίαζαν τις ελευθερίες μας και τα δικαιώματά μας ε, και αυτή η παρέμβαση μπορεί να αποτελεί διακριτική μεταχείριση εναντίον μας. Ε, όμως δεν έχει αναλυφθεί ακόμα δράση. Έχουμε λοιπόν την τελευταία δικτατορία στην Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου. Γιατί δεχόμαστε πιέσεις και δεν μπορούμε να διεξαγάγουμε ε, τις ε, δραστηριότητές μας. Αυτό βέβαια επηρεάζει και τους καταναλωτές, γιατί το κόστος αυτό που μας επιβάλλεται πρέπει να το μετακυλήσουμε βεβαίως στους καταναλωτές. Ε, αυτό επηρεάζει βεβαίω και την απασχόληση, καθώς δεν μπορούμε να βαράξουμε περισσότερη αξία. Το Δημαρχείο λοιπόν παραβιάζει τέσσερα διαφορετικά κεφάλαια της, ε, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, δεν συμμαθείς λοιπόν με το άρθρο 49 ε, της Συνθήκης σε ό,τι αφορά την ε, ελευθερία ε, διεξαγωγής εμπορίου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ότι θέλετε να ανοίξετε ένα εστιατόριο σε ένα εμπορικό κατάστημα σε μια ευρωπαϊκή πόλη. Όμως το Δημαρχείο σας επιβάλλει ε, ποιους θα βάλετε σαν ε, σερβιτόρους, ε, σαν ε, μάγειρες, σας λέει ότι δεν μπορείτε να αποδεχθείτε ρευστοτικές κάρτες κτλ. Ή ότι πρέπει να παρουσιάζετε τα, τα προϊόντα όπως το επιθυμούν. Και ειδικά αν τα υπόλοιπα εστιατόρια στο ίδιο εμπορικό κατάστημα δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, φανταστείτε τι συμβαίνει θα αναγκαστείτε να αυξήσετε τις τιμές ε, των δεσμάτων σας λόγω του κόστους. Θα νιώθετε λοιπόν σαν μια μαριονέτα στα χέρια μιας δικτατορίας. Αποτελεί λοιπόν διακριτική μεταχείριση, γιατί οι υπόλοιποι δεν ε, ε, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες. Και μπορείτε να φανταστείτε ότι ο μάγειρά σα, ο σεφ σα, μπορεί να πάρει τι συνταγέ σα και να πάει σε ένα άλλο εστιατόριο, γιατί δεν είναι δικό σα υπάλληλο, είναι υπάλληλο του Δημαρχείου. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει εδώ αυτή η αδικία και αυτή η δικτατορία. Σκεφτείτε και τα δύο εκατομμύρια κατοίκου τη Σεβίλη που επηρεάζονται από όλη αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Να προσθέσω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος τα εξής. δεν λέμε εδώ ότι πρέπει να καταργήσουμε κανόνες ή κανονισμούς. Όχι. Εμείς κάνουμε μια επίκληση για τους ε, ε καταναλωτές μας, τους καταναλωτές της Ευήλης. Γιατί αναγκάζονται να αγοράσουν ψάρια πιο ακριβά. Γιατί παραβιάζεται δική μας ελευθερία άσκησης εμπορίου δεν γίνεται αυτό το δικαίωμά μας σεβαστό στη Σεβίλη. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος από αυτού. Δεν γίνεται σεβαστό το δικαίωμα. Στη Σεβίλη, αν πουλά ψάρια, δεν έχει τι ίδιε ελευθερίε με του υπόλοιπου ε, εμπόρου ε, τροφίμων στην υπόλοιπη Ισπανία ή στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και στη Μερκασεβίγια, όλοι οι ε, φορεί τη αγορά δεν υπόκεινται σε αυτό το καθεστώ. Επομένως, Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε αυτό το γεγονός, το οποίο όλοι γνωρίζουμε. Ε, υπάρχει το θέμα της ιεραρχίας. Έχουμε τις ε, συνθήκες και το Σύνταγμα της Ισπανίας, ε, που θα πρέπει να, να υπερισχύουν των υπόλοιπων νόμων. Εάν αποσυρθούν όλα αυτά και έχουμε αυτό το βάναυσο καθεστώς στον 21ο αιώνα, ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν. Εμεί θέλουμε να δημιουργήσουμε περαιτέρω απασχόληση. Έτσι έχουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο μπροστά μα. Επομένως, ε, ξέρετε ότι υπήρχε και απόφαση του διαμεσολαβητή για απόσυρση ή για, για ε, τερματισμό αυτής της κατάστασης που δεν έγινε όμως σοβαστή. Και αποφασίστηκε ότι θα έπρεπε ε, να καταργηθεί ένας κανονισμός απολύσεων που θα οδηγούσε στην απώλεια πολλών θέσεων εργασίας. Δεν μπορείτε λοιπόν να μας πείτε ότι μιλάμε εδώ για εσωτερικούς κανόνες εθνικού δικαίου. Όχι, μιλούμε για τους πολίτες μας τον 21ο αιώνα και δεν είμαστε σε θέση να τους ε, παράσχουμε θέσεις εργασίας. Το μόνο που θέλουμε είναι να γίνει σεβαστή αυτή η ελευθερία μας. Ε, σύντομα παρακαλώ, ο κύριος Ραφαήλ Ντομίγκες που είναι ε, πρόεδρος του συνεταιρισμού της ε, Μερκασεβίγια ζήτησε να μιλήσει. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον κύριο Μάιερ που μας επέτρεψε να παρουσιάσουμε και τη δική μας γνώμη επί του προκειμένου θέματος. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να λάβω το λόγο. Το θέμα αυτό αναφέρεται στο άρθρο 49 της Συνθήκης της Λισαβόνας για την ελευθερία εγκατάστασης. Πρέπει να πούμε ότι στη Μέρκα Σεβίγια δεν παραβιάζομαι την ελευθερία αυτή. Και υπάρχουν διακριτικές ε, παραχωρήσεις για όλο το διάστημα λειτουργίας της Μέρκα Σεβίγια. Όταν λοιπόν υπέγραψαν ε, τη σύμβαση, εγνώριζαν τις, τους όρους, τα υπέρ και τα κατά, και τα δέχτηκαν όλα υποχρεώσεις και δικαιώματα. Τώρα, σε σχέση με αυτά που λέγουν για την παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, πρέπει να σας πω ότι προφανώς το δημόσιο αποσκοπεί και έχει πρόθεση να προστατεύει τους καταναλωτές. Εμείς δε τηρούμε όλη την ισπανική νομοθεσία και παρέχομαι δημόσια υπηρεσία για να λειτουργεί η ελεύθερη αγορά και ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Σε αυτά συμβάλλουμε και εμείς. Η αγορά των ηχθείων είναι πιο ανταγωνιστική από κάθε άλλη και ισχύουν καθαρά κριτήρια προσφοράς και ζήτησης εκεί. Αν υπάρχει μεγαλύτερη ε, ποικιλία, πέφτουν οι τιμές για τον καταναλωτή και διαμορφώνονται όπως ελεύθερα, μόνο με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Η Μέρκα Σεβίγια παίρνει ένα ποσοστό ανάλογα με την τιμή των ψαριών. Οπότε υπάρχει ένα παράδοξο εδώ. Αν δεν πουλιέται το προϊόν, η Μέρκα Σεβίγια δεν παίρνει τίποτα, δεν χρεώνει για τις υπηρεσίες που παρέχει. Επίσης υπάρχει και ε, φορολογική διαφάνεια, γιατί η φορολογική απάτη είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Οπότε υπάρχει ανταγωνισμός και πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν. Υπάρχουν λιγότερες ε, επιχειρήσεις λοιπόν. Μία από τις ε, υπηρεσίες που παρέχουμε εμείς είναι ότι ε, παρέχουμε τη δυνατότητα ατομικών πωλήσεων. Πρόσφατα, α, η Μέρκα Σεβίγια είναι μια δημόσια υπηρεσία και διοργανώθηκε και μια εκστρατεία διότι θέλουμε και θέλουμε να υποβάλλουμε μια αναφορά προκειμένου περί της ε, προσφοράς και ποιότητας στους καταναλωτές. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την προσφορά στους πολίτες και να διασφαλίσουμε και την παροχή ποιοτικών προϊόντων. Διεξάγουμε επιθεωρήσεις στην ε, ποιότητα των προϊόντων, θέλουμε ε, ασφάλεια τροφίμων, περιβαλλοντική ασφάλεια και ε, προστασία ε, των ε, προστατευομένων ειδών. Επίσης θέλουμε να καταπολεμούμε τη φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή. Θέλουμε να προστατεύουμε τους καταναλωτές. Αν δεν τα είχαμε όλα αυτά, θα είχαμε λιγότερες επιχειρήσεις στην αγορά, λιγότερη ποικιλία θα είχαμε λιγότερους εμπόρους και οι μεγάλες επιχειρήσεις θα ήλεγχαν την αγορά. Δεν θα είχαμε ε, φορολογική διαφάνεια, θα είχαμε λιγότερη λασιμότητα και φυτογειονομικούς ελέγχους. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε συνολικά είναι να αποφύγουμε καταχρηστικές πρακτικές και βεβαίως δεν θέλουμε να δίνουμε λάθος πληροφορίες και σε εσά. Στην πόλη μας ε, χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ και γίνονται εκστρατείες ε, για το θέμα, αλλά αν δείτε και ε, την έκθεση που έχει καταρτιστεί από τον διαμεσολαβητή θα καταλήξετε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτή είναι μια μη δεσμευτική έκθεση με προτάσεις. Ε, εμείς ε, δεν θέλουμε μονοπωλιακό έλεγχο της αγοράς. Οι δε καταναλωτές της Σεβίλη υπερασπίστηκαν το υπάρχον σύστημα και θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις ε, αν δεχτείτε την πρόταση ε, των άλλων. Ευχαριστώ. Για τις επιτροπές, η κυρία Λεσέν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους της Επιτροπής, όπως υπενθύμησε και ο υπογράφων την αναφορά, πρόκειται για την άσκηση της δραστηριότητας ε, χοντρεμπορίου στην ε, ηχθή αγορά της Σεβίλης. Η υποχρεωτική προσφορά κάποιων υπηρεσιών προς τους χοντρεύωρους κατά κάποια ε, συγκεκριμένη αμοιβής δεν ανταποκρίνεται στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε όσον αφορά την ελεύθερη κατάσταση ούτε όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στην απάντησή μας του Φεβρουαρίου η η Επιτροπή για θέματα ανταγωνισμού αναφέρει ότι δεν μπορεί να πάρει θέση όσον αφορά την υλοποίηση αυτών των κανόνων. Αρμόδια είναι μια εθνική αρχή ανταγωνισμού. Ζητήσαμε λοιπόν από τους αναφέροντες να αποτανθούν στην εθνική αρχή της χώρας τους. Τώρα, όσον αφορά την προσφορά υπηρεσιών έναντι ε, αμοιβή προς τους χονδρεμπόρους, όντως δεν συμβαδίζει με το αντίστοιχο άρθρο της σύμβασης που αφορά την ελεύθερη εγκατάσταση. Η επιβολή υποχρεωτικών υπηρεσιών όπως μεταφοράς, τιμολόγησης, τέτοιου είδους ε, ρυθμίσεις παραβιάζουν την ε, άσκηση της δραστηριότητας των ε, χοντρεμπόρων ιδιαίτερα αυτών που συνήθως προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες στους πελάτες τους. Το κόστος αυτών των υπηρεσιών σαφώς και μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό στοιχείο για τους εμπόρους αυτούς. Δεν αποκλείεται επίσης αυτού του είδους οι περιορισμοί να αντιβαίνουν της ελεύθερης προσφοράς υπηρεσιών στην αγορά ε, αυτή της Μερκασεβίγια. Πρόκειται λοιπόν για περιοριστικούς όρους. Μπορεί κανείς να δικαιολογήσει όμως τα μέτρα αυτά αν ε, μπορεί να επικαλεστεί το δημόσιο συμφέρον. Ζητήσαμε λοιπόν ποιοι είναι οι λόγοι που δικαιολογούν αυτή την ιδιαίτερη ρύθμιση, αυτούς τους ε, κανονισμούς, γιατί εφαρμόζεται μόνο στους χοντρεμπόρους και όχι στους υπόλοιπους. Ε, εμπόρους παρόντες στην αγορά της Σιβίλ ε, και ποια είναι η αναλογικότητα, ποια είναι η διαφάνεια όσον αφορά τις ε, τιμές που επιβάλλονται και αν υπάρχουν άλλοι κανόνες που επιβάλλονται λιγότερο περιοριστικοί, οι οποίοι όμως δεν έχουν ε, επιλεγεί από τις δημοτικές αρχές. Περιμένουμε την απάντηση γιατί θέλουμε να δούμε αν υπάρχει αναλογικότητα και αν υπάρχουν λόγοι που δικαιολογούν την επιλογή αυτών των κανόνων. Ε, ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να στηρίξω την αίτηση των αναφερόντων. Εγώ είμαι από την περιοχή αυτή, γνωρίζω λοιπόν πολύ καλά το θέμα. Πρόκειται για παροχή υπηρεσιών παράνομη που επιβάλλει η περιοχή της ε, Σεβίλης στους χοντρεμπόρους ε, ψαριών. Η Επιτροπή θα στείλει μια επιστολή στις Ισπανικές Αρχές ζητώντας ε, επιπρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές ε, στη Μαρκασεβίλια για να δούμε κατά πόσο αυτό συμμορφώνεται με το άρθρο 49 της ε, συνθήκης. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει την εξέταση των γεγονότων επιτόπου έτσι ώστε να δούμε η απόφαση των Ισπανικών δικαστηρίων εάν επιβεβαιώνεται. Σαν Ευρωβουλευτής από την Ισπανία πιστεύω ότι θα πρέπει να επικαλεστούμε την αρχή του ανταγωνισμού, την προστασία των καταναλωτών και την ελευθερία εγκατάστασης. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που μόλις ακούσαμε από την Επιτροπή, ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, Κανείς δεν ξέρει γιατί συνεχίζουν να επιβάλλονται αυτοί οι κανόνες στους χονδρεμπόρους και όχι σε, άλλες, σε άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε μια συγκεκριμένη απάντηση, να ακούσουμε τα επιχειρήματα όλων, αλλά σε καμία περίπτωση να μην κλείσουμε την υπόθεση. Ε, προφανώς η αναφορά παραμένει ανοιχτή, γιατί αυτή είναι η συνήθις διαδικασία. Η Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι ε, υπάρχει εθνική αρμοδιότητα και όταν πρόκειται για την ε, επιστολή, όταν λάβουμε την απαντητική επιστολή της Ισπανικές Αρχές θα δούμε για το άρθρο 49 και αφού δούμε τι θα πούν οι Ισπανικές Αρχές θα δώσουμε συνέχεια αναλόγως στην αναφορά αυτή. Εγώ είμαι ευρωβουλευτής αλλά ε, ε, ε, είμαι ένας πολίτης του κόσμου δηλαδή και συμφωνώ με αυτά που ακούσαμε. Υπάρχει ένα σύστημα που τροφοδοτεί με προϊόντα τους πολίτες, τους καταναλωτές και υπάρχει και έλεγχος και αυτό είναι καλό πράγμα. Γιατί πρόσφατα είδαμε τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει επιθεώρηση των τροφίμων. Αναφέρομαι στο ε, βακτηρίδιο ε κόλλη και της, ε, την αναταραχή που προκάλεσε στην αγορά. Νομίζω ότι η ασφάλεια και η χνηλασιμότητα, η ανιχνευσιμότητα είναι πολύ σοβαρά θέματα και εκεί πρέπει να υπάρχει δημόσια παρέμβαση. Όταν δεν υπάρχει, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα. Καμιά φορά υπάρχουν προβλήματα και όταν ε, παραγρυπνούμε. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει δημόσιος έλεγχος, χρειάζεται φορολογική διαφάνεια, ε, δημοσιονομική διαφάνεια, γιατί αυτό βοηθάει και τους μικρούς παραγωγού και τους καταναλωτές. Στην Ισπανία Υπάρχουν οι δημόσιοι φορείς που θα πρέπει να κάνουν αυτές τις επιθεωρήσεις. Αυτό δεν συζητείται. Ο δημόσιος χαρακτήρας αυτών των επιθεωρήσεων που διεξάγει η Μέρκα Σεβίγια δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Οι δημόσιες επιθεωρήσεις επιτρέπουν να λειτουργεί καλά η αγορά και να είναι και δίκαιος ο ανταγωνισμός στην αγορά αυτή. Οι καταγγελίες που ακούσαμε από τους χονρεμπόρους είναι αντιφατικές. Οι πωλήσει ηχθείων και η αγορά γενικά στην Σεβιλή είναι πιο ανταγωνιστική από κάθε άλλη αγορά. Είναι μικρότερος όγκος, αλλά είναι και φθηνότερα οι τιμές. Θα πρέπει λοιπόν να σταθμίσουμε τα πράγματα, δηλαδή τα, τα, πράγματα, τα συμφέροντα των παραγωγών με τα συμφέροντα των καταναλωτών. ώστε να έχουμε καλύτερη ε, δημοσιονομική διαφάνεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για πωλήσει. Έτσι λοιπόν υπάρχει ελευθερή αγορά και αν δεν παρενέβαινε το δημόσιο θα δημιουργεί το μονοπόλιο. Λάβετε το υπόψη, ακόμα τα εξετάζουμε και εμείς όλα αυτά, δεν έχουμε αποφασίσει τίποτε, αλλά όταν ακούσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έχουν να πούν οι αρμόδιες αρχές, τότε θα προχωρήσουμε. Και αν η επιχείρηση, ε, αν ε, υποβληθεί αναφορά άλλη, θα δούμε τον κύριο Τουργκάης και μετά κύριε σε εσάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα αρχικά να καλωσορίσω τους συμπατριώτες μου. Η Επιτροπή Επιχειρήσεων, όπως και χονδρέμποροι, πάντα είναι ευπρόσδεκτη στο Κοινοβούλιο. Εγώ γνωρίζω ε, τι συμβαίνει στι αγορέ γιατί συμμετείχα εκεί πέρα στο Συμβούλιο για τον Μπιλμπάο και ήμουν στο αντίστοιχο Συμβούλιο και θυμάμαι αρκετά προβλήματα που είχαμε αντιμετωπίσει ε, εκεί εκείνη την εποχή. Ένας, υπήρχε ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών ε, εκ μέρου των χονδρεμπόρων και είναι γνωστές συμπεριφορέ αυτέ στον Μπιλμπάο και σε άλλε αγορέ, δηλαδή. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι πράγματι ακολούθησα, παρακολούθησα με ενδιαφέρον ε, την συζήτηση, αυτό που είπαν τα δύο μέρη εδώ και θα ήθελα ε, να αναφερθώ στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ήταν αρκετά ξεκάθαρη η άποψή της και όπως είπε και ο συνάδελφος Μιγγέλ, είναι μια πρώτη εξέταση της ε, υπόθεσης. Αυτή η θέση μας επιτρέπει να πούμε ότι περιμένουμε περαιτέρω πληροφορίες. Αν η Επιτροπή λοιπόν πει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ασυμβατότητας με το άρθρο 49 της ε, Συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν κάτι τέτοιο ισχύει, Κυρία Πρόεδρε, αν η Επιτροπή πει ότι περιμένει περαιτέρω πληροφορίες και ότι έχει αμφιβολίες, πρέπει να περιμένουμε την απάντηση μέσω ότου οι ισπανικέ αρχέ ε, αντιδράσουν, δώσουν την απάντησή του και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τον διάλογο με μια δεύτερη εξέταση είτε είναι, θα είναι η συγκεκριμένη αναφορά είτε μια άλλη αναφορά που θα αποβληθεί από κάποιον άλλο Ισπανό πολίτη. Θα ήθελα λοιπόν απλώ να πω ότι η αναφορά αυτή παραμένει ανοιχτή και περιμένουμε περαιτέρω πληροφορίε. Συνάδελφε, κυρία Χιμένες, ζητήσατε σύντομα παρακαλώ γιατί έχουμε πολύ δύο ε, λόγια, γιατί δεν μας μένει πολύ λόγος ακόμα, πολύς χρόνος συγγνώμη. Όλη αυτή η έλεγχη είναι απαραίτητη και αν αυτή η δημοσιονομική διαφάνεια ε, οργανώνεται με έναν καλό τρόπο αλλά ε, εφαρμόζεται μόνο στους χοντρεμπόρους, τότε αυτή η κατάσταση καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο ακατανόητη. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε την εξέταση μέχρι να φτάσουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ε, δεν ξέρω αν ο αναφέρον θα ήθελε. Ένα λεπτό παρακαλώ, ωστόσο, όχι παραπάνω. Ναι, ευχαριστώ. Απλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που μας ε, άκουσε και θέλω να σας πω ότι συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Μέγερ και εγώ είμαι πολίτη του κόσμου. Δεν είμαι μόνος, μόνο πολίτη τη σεβίλη. Ω πολίτης του κόσμου λοιπόν πραγματικά ε, έχω αναστατωθεί και με προβληματίζει ε, τα μάλα αυτή η κατάσταση, γιατί βλέπω ότι στη Σεβίλη εφαρμόζονται κανόνες που δεν ισχύουν για τον υπόλοιπο, του, τον υπόλοιπο κόσμο. Η δημοσιονομική διαφάνεια, ε, η ανιχνευσιμότητα, η υγειονομική έλεγχη, όλα αυτά είναι εντυπωσιακά στοιχεία. Όμως, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάτι το οποίο δεν λειτουργεί καθόλου. Στη Σεβίλη υπάρχουν αυτοί, όλοι αυτοί οι έλεγχοι της δημοσιονομικής διαφάνειας και όλα τα λοιπά, αλλά όλα αυτά ισχύουν μόνο για τους χονδρεμπόρους, τους ηχθιεμπόρους χονδρικής. Ενώ οι υπόλοιποι έμποροι ε, φρούτων, λαχανικών κτλ. δεν υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις. Ε, ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντως ε, δεδομένο ότι η υπόθεση θα παραμείνει ανοιχτή περιμένοντας περισσότερα στοιχεία από τη μεριά της Επιτροπής και επομένως μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Ε, της κυρίας Μπέιτμαν από την Μεγάλη Βρετανία σχετικά με άδικους και κατά όρους τα συμβόλαια μίσθωσης καταστημάτων κατανάλωσης ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχει ε, η κυρία Μπέιτμαν δεν είναι εδώ. Παρακαλώ την Επιτροπή, ε, ε τον κύριο Φερέ, Περέιρα να μας παρουσιάσει το πρόβλημα. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Στο πρώτο μέρος της αναφοράς η αναφέρουσα αναφέρει την εκμεταλλευτική φύση των συμβάσεων μεταξύ εταιριών που είναι ιδιοκτήτες ε, της, ε, του ΠΑΜΠ και των, των μισθωτών. Στο δεύτερο κομμάτι η αναφέρουσα ε, ζητεί νομική αρρωγή για να δώσει συνέχεια το θέμα δικαστικός. Σχετικά με το πρώτο μέρος της αναφοράς, ενώ δεν είναι απόλυτα σαφές αν η αναφέρουσα ε, ε, η αναφορά έχει σχέση με το δίκαιο ανταγωνισμού. Η Κομισιόν το είδε το θέμα και μέσα από αυτό το πρίσμα και σημειώνει η Κομισιόν ότι η αγορά των Βρετανικών pub είναι ανταγωνιστική 45% ε, της αγοράς περίπου ελέγχεται συγκεκριμένα από ελεύθερους υποχρεώσεων εμπόρους που είναι γνωστοί και ως free houses. Αυτή αυτά τα free houses δεν έχουν εμπορική σχέση με τις εταιρείες των pubs. Το υπόλοιπο 55% της αγοράς ελέγχεται από από 8 εταιρείε pub. Η Κομισιόν ήρθε σε επαφή και με την αρμόδια αρχή για τον ανταγωνισμό, το OFT, Office of Fair Trading, στη Βρετανία και έμαθε η Κομισιόν ότι το Office of Fair Trading, η αρχή του ανταγωνισμού, ολοκλήρωσε πρόσφατα μία έρευνα στον τομέα των pub στη Βρετανία και κατέληξε ότι δεν υπάρχουν ε, προβλήματα στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Εις ό,τι αφορά το δεύτερο μέρος της αναφοράς, η Κομισιόν παρέπεμψε την αναφέρουσα στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου για να βρει τη νομική αρρωγή που χρειάζεται η αναφέρουσα από εκεί και να ε, προσφύγει στα δικαστήρια. Ευχαριστώ πολύ νομίζω ότι οι προτάσεις που κάνετε στο κείμενο μοιάζει να είναι πραγματικές. Επομένως, ε, ε, χαίρομαι ιδιαίτερα ότι και σε προσωπικό επίπεδο τη συμβουλεύει για το πού μπορεί να απευθυνθεί προκειμένου να βρει συνηγόρου για να υποστηρίξουν την υπόθεση της στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ε, τελειώσαμε με αυτήν την ε, ε, αναφορά και μιας και ήρθε η πρόεδρος η κυρία Ματσόνη της παραδίδω την έδρα. No, no, no. You have to leave anyway. Okay. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Παλιαδέλη που με αντικατέστησε. Όπως είπα, εκπροσωπούσα σε μία διάσκεψη για το περιβάλλον την Επιτροπή Αναφορών. Πάμε στο σημείο 11 τώρα. Για τις ανακοινώσεις μου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών μετά τη χθεσινοβραδινή συνάντησή τους. Θα τα πω στα γρήγορα. Ε, e Νομίζω ότι έχουν ε, διανεμηθεί σε όλα τα μέλη τα σημεία 1 και 2. Πρόκειται για απόφαση των συντονιστών να συγκεντρώσουν τις ε, αποφάσεις που αφορούν την έκθεση ΟΚΕΝ. Δηλαδή να δούμε πώς μπορούν να κλείσουν οι υποθέσεις αυτές βάσει αυτών που αποφασίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την έκθεση ΟΚΕΝ. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα ιδιοκτησίας, δικαιώματα ιδιοκτησία. Εδώ πάλι κάνουμε μια έκκληση προ την Ισπανική κυβέρνηση που αφορά τον νόμο περιακτών της Ισπανίας. Οι συντονιστές αποφάσισαν να εξετάσουν ε, μια έκθεση πρωτοβουλίας. Αποφασίσαμε επίσης να οργανώσουμε μια ομάδα εργασίας, ένα εργαστήριο εδώ στην Επιτροπή Αναφορών καθότι ο αριθμός των αναφορών με τις οποίες ασχοληθήκαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση ήταν εξαιρετικά αυξημένος. Θεωρούμε επίσης ότι τα δικαιώματα ιδιοκτησίας θα πρέπει να εξεταστούν στα πλαίσια μιας ακρόασης, την οποία οργανώνουμε με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέμα που αφορά άμεσα και τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα οργανωθεί αυτή η ακρόαση στην... την επόμενη μάλλον τον επόμενο Οκτώβριο στις 6 Οκτωβρίου. Θα αναφέρουμε την απόφασή μας στους υπογράφοντες ε, την αναφορά αυτή με επιστολή που θα του σταλεί. Όσον αφορά τώρα την επίσκεψή μας στη Βουλγαρία, το πρόγραμμα είναι ολοκληρωμένο. Επίσης θα επισκεφτούμε και το Βερολίνο. Οι συντονιστές αποφάσισαν να αναβάλουν την επίσκεψη αυτή στο Βερολίνο καθότι δεν μπορούμε να οργανώσουμε αυτή τη στιγμή την επίσκεψη αυτή. Σημείο 4 της ημερησίας διάταξης, προφορική ερώτηση που θέλαμε να υποβάλουμε με την Επιτροπή Αλίας όσον αφορά τα προϊόντα Αλίας. Αποφασίσαμε να αναβάλουμε και αυτήν την προφορική ερώτηση καθότι το ΕΛΚ οργανώνει μια ακρόαση με το θέμα αυτό. Περιμένουμε λοιπόν την ακρόαση αυτή έτσι ώστε να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και να υποβάλουμε μία ακριβέστερη ερώτηση. Σημείο 5. Ο κύριος Κλάιν, υπογράφων την αναφορά που έχει συζητηθεί εδώ πολλές φορές στην Επιτροπή μας, έλαβε μία απάντηση <clears throat> από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που μας οδήγησε στην απόφαση να απευθυνθούμε στον αρμόδιο επίτροπο. Μια ανεπίσημη συνάντηση με τον αρμόδιο επίτροπο πιστεύουμε θα επιτρέψει την επίληψη αυτού του θέματος που θεωρούμε καθοριστικό, εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, μετά από μια δύσκολη διαπραγμάτευση με τον πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, θα προετοιμάσουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ συμφωνεί με το αίτημά μας. Θα προετοιμάσουμε λοιπόν μία έκθεση πρωτοβουλίας για ένα θέμα που μέχρι τώρα είχε, το είχαμε επεξεργαστεί υπό μορφή γνωμοδότησης. Ο συνάδελφος Βαλεάν και λέτε είναι υπεύθυνοι. Από εχθές το βράδυ μέχρι αύριο, έχουμε δηλαδή 48 ώρες, έτσι ώστε να σχολιάσετε την ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε απόφαση εχθές, καθότι το έγγραφο αυτό μοιράστηκε με μεγάλη καθυστέρηση. Έχουμε νομίζω 48 ώρες. Πρέπει σήμερα όλοι να έχετε την ημερήσια διάταξη η οποία θα εγκριθεί μετά από 48 ώρες. Ο συνάδελφος Βίλι Μάγερ έθεσε και το θέμα της αναφοράς των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε χθες και αποφασίσαμε να θέσουμε σαν θέμα συζήτησης την ασφάλεια της ενέργειας κυκλοφορίας ε, στον Ισπανικό ενέργειο χώρο. Ζητήσαμε επίσης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών. Αυτά ήταν τα θέματα που συζητήσαμε χθε ε, μεταξύ συντονιστών. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Δεν έχω άμεση ένσταση. Ερω... Α, ο κύριος, εξ του κυρίου Μπουσουτήλ ζητώ η αναφορά 1073-2010 από Μπ αναφορά να γίνει Α αναφορά. Σε 70, σε 1073 του 2010. για την Ισπανική νομοθεσία για τις ακτές. Καλό είναι να καταλήξουμε σε έκθεση. Είχαμε συμφωνήσει ε, ως συντονιστές να περιμένουμε την απάντηση των Ισπανικών αρχών και μετά να αποφασίσουμε στην Επιτροπή τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα διαδικαστικά. Ε, γιατί Ορισμένοι μπορεί να, ορισμένες ομάδες μπορεί να μην θέλουν να ε, προδικάζουμε με αυτοματισμό τις διαδικασίες. Ακόμα δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ε, και να πούμε 100% ότι θα καταλήξουμε σε έκθεση. Αυτή θα είναι μια διαδικασία. Έχουμε καθορίσει πέντε σημεία, είναι σωστά και ένα είναι σημαντικό ότι θα ζητήσουμε ενημέρωση του Κοινοβουλίου από τις Ισπανικές Αρχές σχετικά με το τι γίνεται με την νομοθεσία αυτή τώρα στην Ισπανία και μετά θα δεσμευτούμε για τη συνέχεια που θα δώσουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή άμεση ένσταση σε αυτά που είπατε, απλώς διευκρινιστικά πρόσθεσα αυτά. Ευχαριστώ. Υπογραμμίσατε το πρώτο σημείο, αυτή δηλαδή, ε, αυτό το αίτημα προς τις Ισπανικές Αρχές ήδη υπάρχει. Επανέρχομαι στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε σημειώσει το αίτημά σα. Ε, περνάμε λοιπόν στο σημείο 14. 11.09 το 2010 τη Σιμών Άιλερ, γερμανική ηθογένεια, σχετικά με την ενίσχυση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση Amici dei Bambini. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην αναφέρουσα. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, λέγομαι Σιμώνε Άιλερ. Πριν από ένα χρόνο, μέσω των ε, γερμανικών ΜΜΕ, διεπίστωσα κάτι συγκλονιστικό. Το λόμπι των υιοθεσιών και τη χρηματοδότησή του μέσα από ενωσιακά κονδύλια. Η Αμίτσι Ντέι Bambini έχει πολύ ε, ισχυρό λόμπι και προσπάθησε να πείσει να ξανανοίξει στις διεθνείς διακρατικές υιοθεσίες η Ρουμανία. Έγιναν πολλές διασκέψεις και πάντοτε παρουσιαζόταν η σημερινή ρουμανική πραγματικότητα. Οι διεθνείς υιοθεσίες αντιμετωπίζουν κρίση. Υποδιπλασιάστηκε σε όλο τον κόσμο μετά την απόφαση της Ρουμανίας η απόφαση αυτή. Πολλές ε, τριτοκοσμικές χώρες τα τελευταία χρόνια σταμάτησαν ή περιόρισαν τις διεθνείς υιοθεσίες ε, ε, λόγω του εμπορίου παιδιών. Η ζημιά που γίνεται ε, είναι περισσότερο γινεται ειναι σαφή στη Ρουμανία. Δεν υπάρχει προστασία των παιδιών, δημιουργείται ελεύθερη αγορά για τα παιδιά. Δεν πρόκειται για το καλό των παιδιών, πρόκειται για τον κορεσμό της ζήτησης για παιδιά και βεβαίως ε, ε, τα λεφτά παίζουν μεγάλο ρόλο. Είναι γνωστό ότι οι υπηρεσίες υιοθεσία ε, αμείβονται για τα παιδιά που παραδίδουν. Πολλές φορές έργα ανταλλάσσονται με παιδιά, κερδοφόρα έργα. Ο Γκίντερ Φερχόιγκεν που ήταν υπεύθυνο για τη διεύρυνση, είπε ότι οι διεθνείς υιοθεσίε είναι νομιμοποιημένο εμπόριο παιδιών. Ε, εγώ εργάστηκα ως εθελόντρια σε ένα κέντρο παιδιών, προστασίας παιδιών και είδα τις συνθήκες ε, διαβίωση σε τέτοια κέντρα των παιδιών. Δεν υποστηρίζονται, δεν προωθούνται ούτε προσπαθούν κανείς να βρει δυνατότητες για να ξαναγυρίσουν στις οικογένειές τους τα παιδιά αυτά. Αντίθετα, σπάζει ε, ο δεσμός με την οικογένεια το νωρίτερο δυνατό. Ο χρόνος παραμονής στο κέντρο είναι ένας χρόνος που επιτρέπει να επιβιώσουν τα παιδιά μέχρι να τα υιοθετήσει κάποιος. Και διαπίστωσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί την Αμίτσι Ντεϊμπαμπίνη η οποία είναι ε, μια υπηρεσία υιοθεσιών. Λένε ότι ε, είναι ένα κίνημα των θετών γονέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν υποστηρίζει μια υπηρεσία υιοθεσιών και ε, υπάρχουν έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ αυτή τη εταιρεία που χρηματοδοτούνται. Υποτίθεται ότι αυτά τα έργα εξυπηρετούν το, την ευημερία και το καλό των παιδιών γενικότερα. Όπως είπαμε όμως οι υπηρεσίες υιοθεσιών χρειάζονται αυτή τη χρηματοδότηση για να εξεύρουν θετές οικογένειες. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά τον διεθνή υποδιπλασιασμό των υιοθεσιών, οι αμίτσιντε οι μπαμπίνοι αυξάνουν συνεχώς τον αριθμό των υιοθεσιών που προωθούν. Επίσης δεν μου πήρε πολύ χρόνο για να μάθω μέσα από το διαδίκτυο ότι οι αμίτσιντε οι μπαμπίνοι είναι ε, σαφώς κατά της ε, ε, προστασίας των παιδιών σε κέντρα και που δεν είδε θέλουν να υπερβαίνει το διάστημα αυτό παραμονής των παιδιών σε κέντρα ε, τη διετία. Ε, Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ένα δίκτυο ε, φίλων του Αμπίνση Βαμπίνη που ε, μεγαλώνει. Αυτά τα έργα δεν αναφέρονται λέει κομισιόν στις διεθνείς υιοθεσίε, αλλά την ε, παρακολούθηση και υποστήριξη των οικογενειών και των παιδιών. Ε, όμως ε, αυτό μπορεί να είναι πραγματικά ε, ένας τρόπος να μπει αλεπού στο κοτέτσι. αυτά που παρατηρούνται στις απαντήσεις είναι ότι πρόκειται για αρμοδιότητα ε, κρατών μελών. Αναρωτιέμαι, αν δεν είναι υπεύθυνη για αυτά τα θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί παρακολουθεί τότε η Κομισιόν την ε, κατάσταση στη Ρουμανία εκ του σύνεγγης. Η Κομισιόν παρατηρεί ε, παραπέρα ότι η Ρουμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ιδιαίτερη θέση. Είναι το μόνο κράτος μέλος που de facto απαγόρευσε τις διεθνείς ιδιακρατικές υιοθεσίες. Όμως ε, για τους αλλοδαπούς είναι επίσης de facto να πάρουν παιδιά από άλλες χώρες, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Ιταλία, τη Γαλλία κλπ. Η Ρουμανία λοιπόν δεν έχει ιδιαίτερη θέση γιατί η Ρουμανία δρά όπως τα παλιά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν εξήγαγαν ε, τα παιδιά τους. Συνοψίζω και επαναλαμβάνω την αναφορά μου αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προωθεί και υποστηρίζει τις υπηρεσίες υιοθεσιών έτσι ε, ε, δίνοντας περισσότερα ενάψματα για τη λειτουργία της αγοράς στον τομέα αυτό. Δεν θα έπρεπε από κοινού να δημιουργηθεί μια δομή που θα προστατεύει τα παιδιά κάθε χώρας προστατεύοντάς τα ε, μέσα στους κόλπους της οικογένειας όπως έγινε στη Ρουμανία ήδη και μάλιστα με αξιοσημείωτη επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος, κύριε Νεγρό, από την οργάνωση Μίτσου Ντεμπαμπίνη είναι εδώ, επομένως μπορούμε να δώσουμε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ονομάζομαι, μιλώ εκ μέρους ε, του, ε, της οργάνωσης αυτής. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι πρόκειται για έναν διαπιστευμένο οργανισμό που βεβαίως και αναλαμβάνει ε, διεθνείς υιοθεσίες, παράλληλα όμως παραμένει μια μη κυβερνητική οργάνωση διαπιστευμένη από την Ιταλική κυβέρνηση ε, με ε, άδεια να ε, προωθεί την προστασία των παιδιών. Έχουμε λοιπόν διάφορες ευθύνες, υποχρεώσεις, δομές για την αποτροπή της εγκατάλειψης παιδιών, αλλά και για την διεθνή συνεργασία. Πριν από δύο εβδομάδες, συζητήσατε ένα σχέδιο το οποίο χρηματοδοτείται ε, και αφορά και τη Ρουμανία. Δύο χρόνια έρευνας ε, χρειάστηκαν ε, για να γίνει αυτό, για να δημορφωθεί ένα σύστημα βαρχής βοήθειας στα παιδιά στη Ρουμανία. Ε, η οργάνωσή μας είναι μια οργάνωση εθελοντική υιοθεσία παιδιών. Δεν λαμβάνουν οι αναδοχοί γονείς, ε, ούτε, ούτε εμείς μάλλον δεν λαμβάνουμε κάποια ε, πληρωμή για τις δραστηριότητε μας. Μπορείτε να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε με αυτό που κάνουμε ή και με τις ε, διεθνείς υιοθεσίε. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε μια μη κυβερνητική οργάνωση που μπορεί να, κάνει, ε, να έχει και άλλε δραστηριότητε και να λαμβάνει ε, χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να χρηματοδοτήσει άλλε δραστηριότητε που δεν έχουν καμία σχέση με τι διεθνεί υιοθεσίε. Εμεί ε, επίση δραστηριοποιούμαστε στον τομέα τη πρόληψη και τη περίθαλψη. Και αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των παιδιών. Εκ μέρους του Προέδρου Μάρκο Γραφίνη θα ήθελα να πω ότι στην Ιταλία η αναφορά αυτή ε, έχει τύχει πολλών κατηγοριών. Αναγκαστήκαμε να πάμε στα δικαστήρια για να την ε, για αυτό την υπόθεση. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Θεωρούμε ότι πρόκειται για σπήλωση του ονόματος της οργανωσής μας και είναι ε, λάθος να συμβαίνει αυτό. Εμείς εργαζόμαστε για την προστασία των παιδιών και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες και στη Ρουμανία όπου ε, εξακολουθούμε να έχουμε εταίρους. Ε, έχουμε εταιρικές σχέσεις με τις τοπικές αρχές στη Ρουμανία. ενδεχομένως να μην συμφωνείτε, αλλά εμείς ε, πιστεύουμε ότι θα, θα έπρεπε να είναι δυνατή ε, η διεθνής υιοθεσία. Όμως, οποιαδήποτε χρηματοδότηση λαμβάνουμε πηγαίνει σε άλλες δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την Επιτροπή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για μία αναφορά που αφορά την συγχρηματοδότηση μιας ε, Ιταλικής ε, οργάνωσης Αμήτρη Δημαμπίνη και θα πρέπει να δικαιολογήσουμε την δαπάνη κοινοτικών κονδυλίων από αυτήν, την, αυτόν τον οργανισμό. Η συγχρηματοδότηση γίνεται μέσω πολλών κοινοτικών προγραμμάτων από το 2001 ως το 2009, από το Europe Aid, FAR, κοινωνικό για την αποφύγη του κοινωνικού αποκλεισμού. Διάφορα δηλαδή προγράμματα κοινοτικά χρηματοδότησαν ε, αυτόν τον ε, Ιταλικό οργανισμό. Πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική ένωση. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι πληρούνται τα κριτήρια από μέρος ε, του οργανισμού αυτού και γνωρίζουμε την ίδια ώρα ότι η Αμίτσι Ντεμπαμπίνη είναι αναγνωρισμένη και Βάσει της συνθήκης της Χάγης, εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα των διεθνών υιοθεσιών. Τα κράτη-μέλη μπορούν λοιπόν να δώσουν, αν θέλετε, την αναγνώρισή τους, τη διαπίστευσή τους σε κάποιους ε, οργανισμούς έτσι ώστε να παίξουν ένα ρόλο σε αυτήν την διεθνή υιοθεσία, σε αυτή τη δραστηριότητα διεθνών ε, υιοθεσιών. Πρόκειται για ενώσεις, πρόκειται για μη κυβερνητικούς οργανισμούς που κανονικά παίζουν ε, ένα συγκεκριμένο ρόλο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο, κυβερνητικός, ο μη κυβερνητικός αυτός οργανισμός έχει ε, αποδείξει ότι πληρεί τα κριτήρια για να συμμετάσχει σε αυτήν την χρηματοδότηση. Τα κονδύλια εδόθησαν για την προστασία παιδιών σε διάφορους τομείς. Έχουν παραδείγματο χάρη προγράμματα για την αποφυγή παράνομων υιοθεσιών, ε, παράνομης εμπορίας παιδιών στην Αλβανία, περίθαλψη παιδιών. Επίσης ε, την πρόθεση βέλτιστων ε, πρακτικών, δικαιώματα των παιδιών για ένα οικογενειακό περιβάλλον, περίθαλψη οικογενειακή για τα παιδιά, υγειονομική περίθαλψη κτλ. Η Επιτροπή επιλέγει κάποια από αυτά τα προγράμματα ελέγχοντας τα κριτήρια Βάσει των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αξιολογούμε το περιεχόμενο των προγραμμάτων, τους στόχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι τα προγράμματα αυτά που συγχρηματοδοτούνται αντιβαίνουν ε, τα δικαιώματα του παιδιού ή κάποια άλλη διεθνή σύμβαση και θεωρούμε ότι ο στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η κοινωνική συνοχή, η ενσωμάτωση των παιδιών σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, παιδική προστασία, περίθαλψη, στήριξη των οικογενειών που έχουν υιοθετήσει παιδιά. Και βεβαίως όλα αυτά συμβαδίζουν με τους στόχους ε, της ε, σύμβασης. Δεν βλέπουμε λοιπόν απολύτως καμία αντίφαση με τους στόχους αυτών των προγραμμάτων. Η χρηματοδότηση η κοινοτική χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό και τους στόχους του κανονισμού. Δεν έχουμε λοιπόν σήμερα απολύτως κανένα λόγο να συνεχίσουμε την εξέταση αυτή την αναφορά. Ευχαριστώ. Η κυρία Ανώκα, έχετε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη υπόθεση, γιατί συνήθως έχουμε απάντηση της Επιτροπής ε, βάσει της ε, αρχής επικουρικότητας. Η Επιτροπή λέει ότι πρόκειται για πλήρη αρμοδιότητα των ε, κρατών μελών και δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αυτό μας λένε πάντα. Βεβαίως και η νομοθεσία αποτελεί ε, πλήρη αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το ερώτημά μου απέναντι στην Επιτροπή είναι το εξή. Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν στην, που αποσκοπούν στην ε, ε, μεταβολή, μεταβολή της νομοθεσίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιβαίνουν στην αρχή της επικουρικότητας. Ιδίως εφόσον αυτές οι δραστηριότητες ε, αναλαμβάνονται από ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται ε, από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τελικά δεν κατάλαβα και θα ήθελα να ακούσω ξεκάθαρα και συγκεκριμένα αυτές οι δραστηριότητες ε, στη Ρουμανία από ποιον χρηματοδοτούνται και για ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες. Ποιο είναι το υπόβαθρο, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει ε, αντίφαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι αυτή η αναφορά από την Γερμανία θέτει επιτάπητος ε, κάτι προφανές. Πρώτον, πρόκειται για ζήτημα επικουρικότητας, το οποίο ε, έχει αναφερθεί πολλές φορές ε, και το έχει εξετάσει αυτό το ζήτημα πολλές φορές η Επιτροπή σε προηγούμενε απαντήσεις τη. Δεύτερον, η σημερινή απάντηση της Επιτροπής επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας για τα ε, διαφορετικά σταθμά, αν θέλετε, ε, που, ακολουθεί η Επιτροπή. Σε άλλα ζητήματα λέει ότι πρόκειται για ζήτημα απεικορικότητα. ταυτόχρονα όμως η Επιτροπή ε, χρηματοδοτεί μία μη κυβερνητική οργάνωση ε, Υπονομεύοντα έτσι την αρχή της επικουρικότητας. Κάτι που είναι απαράδεκτο. Και θα ήθελα να επαναλάβω κάτι το οποίο την προηγούμενη φορά ε, τρεις συντονιστές ε, διαφώνησαν μαζί μου, ε, συγγνώμη, με αυτή την υπόθεση, από μένα την κυρία Βιπή και τον άλλον συντονιστή. Και στη δική μας επιστολή η ε, ε, Επιτροπή απάντησε με έναν ιδιαίτερα δύναμο τρόπο. το τώρα λοιπόν τη συγκεκριμένη υπόθεση, έχουμε μία μη κυβερνητική οργάνωση που έχει έναν τριπλό ρόλο. Ε, με ιδιαίτερες, ιδιαίτερες αντικρουόμενες δραστηριότητε, αν θέλετε. Αρχικά, προωθούν και προασπίζονται τα δικαιώματα των παιδιών. Πολύ καλό και θεμητό. Δεύτερον, εφαρμόζουν τη νέα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ε, υιοθεσίε παιδιών και τις διεθνείς υιοθεσίε παιδιών και τρίτον ασκούν και αυτή την δραστηριότητα της υιοθεσία παιδιών. Φανταστείτε οι συνάδελφοι μέσα σε, ε, ένα τραπεζική υπάλληλοι ταυτόχρονα να είναι να βρίσκονται σε έναν οίκο αξιολόγηση, σε ένα ρυθμιστικό όργανο και σε μια τράπεζα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που σας δίνω. Είναι ο καλύτερος τρόπος να ε, περιγράψουμε και να ορίσουμε την, ε, ε, την ύπαρξη αντικρουόμενων συμφερόντων. Γι' αυτό συμβαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτή τη οργάνωση. Έχουν λοιπόν ένα τερβλό ρόλο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόλυτη ψυχαρήμια μα λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα έπρεπε να είναι απολύτω αποδεκτό. Εγώ όμω δεν μπορώ να αποδεχθώ την ιδέα ότι ο Ευρωπαίος φορολογούμενος ε, και τα χρήματά του μάλλον ε, ε, κατευθύνονται προς αυτές τις δραστηριότητες. Και έχω ένα ερώτημα. Ποια, πώς είναι αυτά τα χρήματα που ε, λαμβάνουν πόσα χρήματα ε, κατευθύνονται προς, την, ε, προς τις διεθνείς υιοθεσίες, για, πόσα για την βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των παιδιών αυτών και πόσα παιδιά έχουν τύχη διεθνούς υιοθεσίας. Πόσα από τη Ρουμανία, πόσα από τη Βουλγαρία ενδεχομένω ή από άλλες χώρες. Γιατί αν κοιτάξουμε τα κονδύλια που, ε, που δίνονται σε μία χώρα και τον, και τον αριθμό των παιδιών που υιοθετούνται σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να υπάρχει ένας συσχετισμός. Πρέπει κάτι να μας πει λοιπόν η Επιτροπή. Ε, αλλιώς θα είναι σαν ε, απλώς να, να αφήνει το καθένα να κάνει ό,τι θέλει και αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Τελευταία μου παρατήρηση Έχουμε εδώ κάτι ενδιαφέρον. Έχουμε μία αναφέρουσα που ήρθε εδώ στην Επιτροπή μας για να παρουσιάσει την αναφορά της. Ωραία. Ταυτόχρονα όμως είχαμε και κάτι ε, πρωτοφανέ, ένα αντιάτορο της Άλτερα κάτι που δεν μπορώ να αποδεχθώ. Κανείς δεν μπορεί βεβαίως να κατηγορήσει την αναφέρουσα, ούτε μπορούμε να κατηγορήσουμε και μια μη κυβερνητική οργάνωση. Δεν θα πρέπει να γίνει παραδεκτό όμως και δεν θα πρέπει να ε, επαναληφθεί στο μέλλον. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι λίγο πιο αντικειμενική ε, ε, και δεν γίνεται να έχει διαφορετικές αντιδράσεις σε διαφορετικές υποθέσεις. Υπάρχει εδώ πέρα σύγκρουση συμφερόντων. Πρέπει να αποφασίσει υπάρχει ή όχι. Εάν υπάρχει, τουλάχιστον να τα ξεκαθαρίσουμε τις νομικές και οικονομικές πτυχές και αυτό να επηρεάσει και την εφαρμογή της διαδικασίας. Και κλείνω εδώ κύριε Πρόεδρε. Να σας υπενθυμίσω συνάδελφοι, ότι η οργάνωση Amici Dei Bambini και άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις είχαν, ε, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό ε, σε lobbying στο Κοινοβούλιο για το ίδιο ζήτημα και στη Ρουμανία και για άλλες χώρες για το ίδιο ζήτημα. Και τώρα με τους νέους κανόνες ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελα αυτή η διαδικασία να σταματήσει. Και ο, ο του Κοινοβουλίου και ο Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου να χειριστούν αυτή την υπόθεση με τα νέα πρότυπα, ε, ηθικά πρότυπα που χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Άλλες παρεμβάσεις υπάρχουν. Όχι. Η αναφέρουσα θέλει να απαντήσει. Η Επιτροπή θα απαντήσει στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Έχετε το λόγο. Η Επιτροπή πρώτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις των ε, αξιότιμων βουλευτών. Βεβαίως, μπορούμε να υποβάλουμε περαιτέρω παρατηρήσεις και στοιχεία για τα συγκεκριμένα πρόγραμμα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και γραπτός. Μπορούμε να σας δώσουμε όλες τις εγκρίσεις ε, για κονδύλια και για χρηματοδότηση που έχουν περάσει από την Επιτροπή. Συγκεκριμένα μπορώ να σας πω για τα προγράμματα αυτά που αφορούν τη Ρουμανία, σε ποιο σημείο εντοπίζονται, για το 2009 παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα Progress, κοινωνικό πρόγραμμα, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 450.000. Πρόκειται για υπηρεσίες κοινωνικές και κάποια διαμεσολάβηση, ερευνητική επίσης δραστηριότητα αλλά και δυνατότητα για τους εμπλεκόμενους φορείς να ανταλλάξουν απόψεις. Έχουμε εξάλλου και τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος. Επίσης, ένα άλλο πρόγραμμα το 2008 θεμελιώδη δικαιώματα πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την δικαιοσύνη οικογενειακή περίθαλψη 430.000 χρηματοδότηση καλύπτει Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία ε. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να υπάρξουν δηλαδή 400 τέτοιες ενώσεις μη κυβερνητικοί οργανισμοί με σκοπό την περίθαλψη και την πρόθεση των ε, αναδόχων. Πρόκειται για μια χρηματοδότηση που έγινε στα πλαίσια του ΦΑΡ με 470.000, ένα άλλο πρόγραμμα Ιταλία-Ρουμανία με σκοπό τη διοργάνωση περιφερειακών ε, συναντήσεων που αφορούν ε, τα παιδιά και την κατάσταση που επικρατεί σε περιοχές αυτές. Αλλά όλα αυτά θα σας τα δώσουμε και γραπτός. Ευχαριστώ. Ρωτήσατε επίσης για την πτυχή της ε, επικουρικότητας, πολιτική οθεσίας. Όντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λάβει μέτρα, δεν υπάρχουν κανονισμοί. Όντως λοιπόν πρόκειται για θέμα που αφορά την εθνική νομοθεσία, την εθνική αρμοδιότητα και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται εδώ τις επιλογές των κρατών. Το επαναλαμβάνουμε αυτό, σεβόμαστε τις επιλογές των κρατών μελών όσον αφορά θέματα υιοθεσία. Και βεβαίως ε, όλα τα κράτη-μέλη έχουν υπογράψει την Σύμβαση για τη Διεθνή ε, Υιοθεσία. Το θέμα των αντικρουόμενων συμφερόντων. Όπως είπα και στην πρώτη μου παρέμβαση, θελήσαμε να αποσαφηνίσουμε το θέμα της χρηματοδότησης. Εμείς δηλαδή κοιτάμε το θέμα αυτό υπό την πτυχή της χρηματοδότησης. Δεν έχουμε λόγο να επικαλεστούμε εδώ αντικρουόμενα συμφέροντα όσον αφορά τουλάχιστον τα κονδύλια και τη χρηματοδότηση. Πρόκειται για μια μη κυβερνητική οργάνωση και θεωρούμε ότι είναι νόμιμη, λειτουργεί στα πλαίσια της Ιταλικής νομοθεσίας, είναι αναγνωρισμένη στην Ιταλία Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι μπορούμε να επιλέξουμε ένα μη κυβερνητικό οργανισμό στα πλαίσια ενός ε, ε, κράτους που ζητά χρηματοδότηση. Τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούμε επίσης θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ε, ζητηθεί από τους οργανισμούς που ζητούν οι οποίοι πληρώνουν τα κριτήρια. Ευχαριστώ πολύ. Η αναφέρουσα έχει το λόγο. Δεν παρακολουθώ και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται κατανοητό το αυτονόητο. Πρόκειται για υπηρεσία υιοθεσιών εδώ και τα έργα που προβάλλει αφορούν την πρόνοια των παιδιών ενώ ο στόχος δεν είναι άλλος από την υιοθεσία. Η απάντηση της Κομισιόν είναι ανεπαρκής και δεν υπησύλθε στην αναφορά μου λεπτομερώς. Επειδή είναι εγκεκριμένη οργάνωση δεν σημαίνει ότι θα υποστηρίζεται ε, άκρητα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω αυτά που ελέγχθησαν ε, μετά από την Κομισιόν. Ούτως ή άλλως θα μας δώσει έγγραφο σημείωμα λεπτομερές η Κομισιόν σχετικά με τη χρηματοδότηση. Οπότε αφήνουμε ανοιχτή την αναφορά μέχρι να υποβληθούν οι πληροφορίες αυτές και θα δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. πρέπει να περιμένουμε μέχρι να λάβουμε όλες τις πληροφορίες και τότε θα δώσουμε απάντηση στην αναφέρουσα. Μπορεί να μπούμε σε θέματα ουσίας εδώ αργότερα. Ε, προχωρούμε λοιπόν στο επόμενο σημείο μας στην ημερήσια διάταξη που είναι το υπαριθμόν 17 αναφορά του Τζον Doherty εξ ονόματος της Irish Drivers Association, ε, Ένωση Ιρλανδών Οδηγών. Θα δώσω το λόγο στον αναφέροντα. Παρακαλώ κύριε. Καλημέρα, λέγομαι John Doherty και είμαι αναπληρωτής πρόεδρος της Irish Drivers Association Στις 8 Ιουνίου του 1972 εμείς ε, ε, οι πολίτες της Ιρλανδίας ε, δεχθήκαμε στα πλαίσια της ένταξης στην Ένωση μια παρέκκληση υπέρ της Ιρλανδίας βάσει άρθρου 14 που θα εφαρμοζόταν από το 82 και αφορούσε στα τελωνιακά τέλη βάσει του άρθρου 25 της Συνθήκης της Ρώμης. Το άρθρο 25 προβλέπει ότι οι τελωνιακοί δασμοί ε, ρυθμίζονται ε, για τα κράτη-μέλη ε, είχε αναφερθεί τότε ότι παραβιάζεται άρθρο του Ιρλανδικού Συντάγματος και γι' αυτό χορηγήθηκε η παρέκκληση, η εξαίρεση. Ε, Επίση έγινε τα αναφορά στο άρθρο 39 της ελεύθερης διακίνησης ε, των εμπορευμάτων ε, στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να τεθεί τέλος της διακρίσης. Επίσης ε, συζητήθηκε το άρθρο 110 πρώην 90 για την προστασία των ε, τοπικών προϊόντων. Η Ιρλανδία δεν πληρεί ε, τα κριτήρια που προβλέπει το άρθρο γιατί δεν ε, κατασκευάζει συναρμολογή μηχανοκίνητα οχήματα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, μέσα από αυτό το πρίσμα το θέμα των εσόδων και την προστιθέμενη αξία ε, στην αγορά. Ε, ε, υπάρχουν ρυθμίσεις και για εισαγόμενα είδη. Ο ΦΥΠΙΑ αλλά και το, το, είναι υψηλό, αλλά και το τέλος ταξινόμησης ανέρχεται στο 36% το VRT το τέλος ταξινόμησης. 73% ε, είναι το σύνολο των φόρων, φόροι επιφόρων. Έτσι λοιπόν, ε, προβλέπεται δε η κατάσχεση του οχήματος αν δεν πληρωθεί το τέλος και επιβάλλεται και πρόστιμο που ανέρχεται μέχρι και σε 10% σύνολο φόρων 83% ε, αυτό παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Ε, επίσης μπορεί να επιβληθεί και από δικαστικά πρόστιμο μέχρι και 5.000 ευρώ. Εμείς θέλουμε να μας δοθεί η δυνατότητα να λάβουμε μέτρα για να σταματήσει η επιβολή αυτού του τέλους ταξινόμησης που είναι τόσο υψηλό και υπάρχουν ε, σχετικές πράξεις για να στηριχθούμε. Οι ε, Βρυξέλλες ήδη έχουν ε, επιβάλει πρόστιμα στα πλαίσια διαδικασίας επί παραβάση κατά της Ιρλανδίας. Θέλουμε λοιπόν να, ε, σε, σε αυτό το θέμα να ε, έχουμε ένα ύψος τέλους εναρμονισμένο με τις άλλες χώρες. Hi, uh, my name is John I'm... Το όνομά μου είναι John και είμαι πρόεδρος ε, της ε, Ανασύσης των Οδηγών. Όσον αφορά αυτό το τέλος ταξινόμησης που ονομάζουμε VAT, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη χώρα μας. Γιατί έχουμε στο σύνταγμά μας την διάταξη που στο άρθρο 38 του συντάγματό μας αναφέρει ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επικαλεστούμε αυτές τις διαδικασίες. Το άρθρο 43 που διέπει θέματα ιδιωτικής ε, ε, ιδιοκτησίας, συγγνώμη, δεν μπορεί να ψηφίζονται νόμοι και διατάξεις που να παραβιάζουν το, το άρθρο αυτό του συντάγματος. Και εδώ υπάρχει σαφής παραβίαση και δεν τηρείται και η αρχή της αναλογικότητας. Πρόκειται για ένα τέλος που πραγματικά ξεπερνάει αυτήν την αρχή και εδώ και τόσα χρόνια πληρώνουμε ένα φόρο που αντιβαίνει των αρχών της εσωτερικής αγοράς. Και όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των ε, αγαθών και των ανθρώπων, και αυτή η αρχή παραβιάζεται. Ζητούμε λοιπόν από την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά το θέμα αυτό σήμερα και θα θέλαμε να έχουμε μια δίκαιη απόφαση, αμερόλεπτη. Θα δώσω όμως το λόγο και στον συνάδελφο. Χωρίς μικρόφωνο. Okay. You're on. This, contentious tax, it comes αυτό το επίμαχο θέμα καλύπτει τη δημοσιονομική πράξη του 92 και τους ειδικούς φόρους. Πρόκειται για το τμήμα 132 και ε, αναφέρεται και αυτό το είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών τότε ε, ε, επιπροσθέτως προς, άλλους, προς άλλα τέλη που μπορεί να χρεώνονται με βάση τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού και με βάση τους σχετικούς κανονισμούς από το 1993 1 Ιανουαρίου ε, θα εισάγεται το τέλος ταξινόμησης οχήματος που θα χρεώνονται, θα επιβάλλονται, θα, καταλάβω, θα καταβάλλονται ε, με βάση τους προβλεπόμενους ε, όρους και συνθήκες βάση του, του άρθρου αυτού. Αυτό είναι ειδικό φόρος και, που εισάγεται από την πίσω πόρτα. Ε, τι είναι τέλος και τι είναι ε, φόρος. Θα πρέπει να εξετάσει το Κοινοβούλιο παρακαλώ το θέμα, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πιστεύουμε ότι εδώ ε, υπάρχει παραβίαση της ελεύθερης διακίνησης. Ιδιαίτερα ε, μεταξύ, ε, υπάρχει πρόβλημα μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και ε, Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Εξετάστε το θέμα. Ξέρω ότι έχει αρχίσει να το εξετάζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει μετά από τις έρευνες που θα γίνουν να ληφθεί σχετική απόφαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τους τρεις. Το λόγο έχει η Επιτροπή. Yes. Uh, so the uh, petitioner... Ευχαριστώ. Ναι, οι αναφέροντες ε, ισχυρίζονται ότι απαγορεύεται αυτός ε, ο τελωνικός δασμός και, θα και ότι μάλιστα είναι και πολύ ψηλός. Δυστυχώς ε, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την φορολόγηση οχημάτων είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Ε, και δεν ε, βρίσκεται στο ύψο των περιστάσεων, αν θέλετε, για να την ύπαρξη μία ενιαία αγορά. Όμω οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να επέλθει μόνο με, ομόφωνη γνώμη, με σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών. Και είναι δύσκολο να αλλάξει η κατάσταση ευρεχηπρόθεσμα. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν προς το παρόν να εφαρμόζουν διαφορετικά καθεστώτα φορολόγηση των αχημάτων ε, στην επικράτειά τους και αρκετά μεγάλο αριθμό κρατών μελών πράγματι ε, επιβάλλουν τέτοιου φόρου. Θα πρέπει βέβαια να γίνεται σεβαστό το άρθρο 110 ε, της συνθήκης ε, που απαγορεύει την ε, διακριτική φορολόγηση άμεσα ή έμεσα σε βάρος προερχόμενα προερχόμενων από άλλα Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, ορισμένες πτυχίες του VRT ε, πράγματι εντάσσεται στο πλαίσιο ε, συνεχιζόμενης διαδικασίας υπό όμως αυτό δεν αφορά το δικαίωμα φορολόγησης, ε, αφορά συγκεκριμένε λεπτομέρειες που παραμένουν σε αυτή τη διαδικασία υπό και για λόγους εμπιστευτικότητας δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Σας διαβεβαιώ όμως ότι δεν συνδέεται με αυτή την υπόθεση. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή έχει ε, προσπαθήσει επισταμένως να ε, άρει τα εναπομείναντα ε, φορολογικά εμπόδια. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι δυνατόν. Δεν έχει καταστεί δυνατόν μάλλον γιατί δεν έχει υποστηριχθεί αρκετά από τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα το 2005 υπήρξε πρόταση οδηγίας αλλά δεν έχει οθετηθεί. σχετικά με το υψηλό φορολογικό συντελεστή και τις κατασχέσεις ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να επιβάλλουν το φόρου όσους φόρους θέλουν αρκεί να μην υπάρχει διάκριση ανάμεσα στα εγχώρια αυτοκίνητα και στα ε, αυτοκίνητα που έρχονται από το εξωτερικό. Και ε, η κατάσχεση είναι ένας τρόπος επιβολής του νόμου αν δεν, αν δεν αποπληρωθεί ο φόρος. Η Επιτροπή βεβαίω μπορεί να εξετάσει περαιτέρω αυτή την αναφορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το συνα... στη συνάδελφο το λόγο. Εγώ δεν θα αμφισβητήσω το γεγονός ότι έχουν δικαίωμα τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν ε, τους φόρους τους. Αυτό είναι μια αρχή την οποία τη δεχόμαστε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει εδώ ένα θέμα ευρωπαϊκό, σημαντικό θέμα, εάν δηλαδή σε μια περιοχή με πολλές ε, συναλλαγές, μετακινήσεις από τη μία και την άλλη πλευρά των συνόρων για συνοριακές ε, εμπορικές ε, συναλλαγές και κυκλοφορία. Πρόκειται για μια περιοχή η οποία είναι περικυκλωμένη από το άλλο κράτος μέλος. Μόνο 7 χιλιόμετρα ουσιαστικά εφάπτεται με το υπόλοιπο ε, Ιρλανδικό κράτος. Πώς ερμηνεύει λοιπόν εδώ η Ιρλανδική κυβέρνηση την επιβολή αυτού του φόρου και πώς τον υπολογίζει κάποιος αγοράζει ένα αυτοκίνητο, παραδείγματος χάρη, στην άλλη πλευρά των συνόρων και το φέρνει και όταν θέλει να καταχωρήσει στα μητρώα της χώρας του αυτό το αυτοκίνητο, ο φόρος που επιβάλλεται ξεπερνάει και τη διαφορά τιμής. Δεν πρόκειται λοιπόν για μία απλή εμπορική, αν θέλετε, αντιστάθμιση. Σε καμία περίπτωση λοιπόν ε, δεν μπορούμε να μην εξετάσουμε το θέμα αυτό. Υπάρχει μια αντίσταση όσον αφορά την πληρωμή αυτού του φόρου. Υπήρξαν κατασχέσεις. Και πολύ σύντομα βλέπουμε ότι κάποιος αν δεν ε, πληρώσει το φόρο Υπάρχουν και μέχρι και ποινικέ ε, διαδικασίες, όχι απλώς δηλαδή έρχεται κάποιος στο σπίτι του και μπορεί να υπάρξει κατάσχεση άμεση, είτε τον σταματάνε στον δρόμο για έλεγχο και του κατάσχουν το όχημα. Σαφώς λοιπόν και πρόκειται για αρμοδιότητα του κράτους μέλους, αλλά πρόκειται και ένα θέμα εμπορίου διασυνοριακού, καθημερινής, αν θέλετε, κυκλοφορίας σε μια περιοχή μεταξύ δύο κρατών μελών που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Γιάρ. Εδώ υποτίθεται ότι τηρεί την νομοθεσία, αλλά οι προθέσεις είναι διαφορετικές. Ε, φόρος ταξινόμησης 36% τι σημαίνει. Σημαίνει ότι διώχνουμε τα αυτοκίνητα από την αγορά μας. Αυτό δείχνει, είναι προστατευτική πολιτική. Απλώς σε ωραία συσκευασία. Μπορούμε να τα πούμε ωραία, να, τα, να λέμε άλλα, αλλά να εννοούμε άλλα. Όταν έχουμε 100 ή 200 ευρώ το φόρο, υπάρχει... Ε, στη Γερμανία τι θα γινόταν αν κάναμε εισαγωγή τέτοιων οχημάτων. Θα έπρεπε να περάσουν το τύφ, θα έπρεπε να αποδείξουν ότι είναι ασφαλή τα οχήματα για δύο χρόνια, να το δηλώσουν κάπου, πληρώνοντας 100-200 ευρώ, λογικό ποσό και είναι και εθνική νομοθεσία. Αλλά 36% αυτό είναι τελείως δυσανάλογο. Και βλέπω ότι η Κομισιόν συμμερίζεται τις ανησυχίες και επιφυλάξεις αυτές. Ε, το διατυπώνει προσεκτικά, αλλά βλέπω ότι ε, ε, δέχεται ότι είναι λίγο ε, ανέδει αν θέλετε να χρησιμοποιούνται οι νόμοι με τέτοιο σκοπό απότερο. Ε, εμείς ε, θέλουμε την ε, ελεύθερη εσωτερική αγορά, είναι πλεονέκτημα ότι την έχουμε, άρα απευθύνω έκκληση στα κράτη-μέλη να μην κάνουν τέτοια φορολογικά κόλπα για να κάνουν προστατευτική πολιτική. Αυτό η Ιρλανδία το κάνει βέβαια γιατί είναι νησί. Ε, αλλιώς θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να το κάνει διότι ε, και ξένες εταιρείες θα ε, διαμαρτύρονταν. Ε, είναι λάθος λοιπόν αυτή η πρακτική. Εμείς όμως τώρα τι θα κάνουμε. Μέχρι τώρα από ό,τι φαίνεται η Ιρλανδία κοφεύει στις φιλικές παρενέσεις της Κομισιόν και η Κομισιόν έχει επιφυλάξεις όπως είπαμε και διαβουλεύεται με την Ιρλανδία. Η Ιρλανδία όμω λέει αυτό είναι δικό μου δικαίωμα, εγώ το βλέπω διαφορετικά και παρακαλώ την Κομισιόν να εξετάσει και κάτι άλλο. Υπάρχει παντού η αρχή ότι ναι υπάρχουν ίδιε αρμοδιότητε εθνικέ, αλλά υπάρχει και ο προσήκον χαρακτήρα των μέτρων και ο αναλογικό χαρακτήρα των μέτρων που εδώ υπερβαίνεται κατά πολύ. Όπω είπα πρόκειται για προστατευτική πολιτική η οποία δεν συμβιβάζεται με του κανόνε της ελεύθερης εσωτερικής αγοράς. Συμφωνώ με τις επιφυλάξεις. Τι θα κάνουμε. Μπορούμε να συντάξουμε και εμεί επιστολή. Θα πρέπει να αποφανθεί η Κομισιόν, γιατί η Κομισιόν στην αναπάντηση λέει ότι από το 2005 ήδη προσπαθεί μέσα από πρόταση οδηγίας να λύσει το πρόβλημα αυτό και η Ιρλανδία εξακολουθεί να αρνείται. Το θέμα είναι τι άλλο μπορεί να γίνει επίσης. γιατί ε, έχουμε εδώ κάποια μηχανία. Παρακολουθούμε αμήχανα και ελαφρώς εκνευρισμένα, για να το πω έτσι ήπια. Μπορούμε να το συζητήσουμε ευρέως το θέμα, αλλά αν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις, τότε δεν θα λειτουργεί και η εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Ναι, καταλαβαίνω. Σε αυτό το σημείο Ας δώσουμε το λόγο μόνο σε έναν από τους τρεις αναφέροντας για μια απάντηση. Και μετά θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε ως Επιτροπή. Actually, Ουσιαστικά κάτι δεν απαντήσατε, δεν καταλάβατε. Εάν κάποιος εισάγει ένα όχημα, η ταξινόμηση είναι 50 ευρώ. Όμως, ένα ΙΧ είναι 3.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το τέλος ταξινόμηση είναι ουσιαστικά τελωνιακός δεσμός. Γιατί το εμπορικό όχημα πληρώνει τόσο λιγότερο, τόσο χαμηλότερο ποσό. Χάσαμε λοιπόν χιλιάδες θέσεις απασχόλησης και ουσιαστικά πρόκειται για μία η εισαγωγή που γίνεται μεταξύ της Δημοκρατίας Ιρλανδίας και της Βόλειας Ιρλανδίας που γίνεται παράνομα, επαναλαμβάνω, είναι αντίθετο με το σύνταγμα της ναι. χώρας. Και δεν δίνονται αυτά τα ποσά στους πολίτες, απλώς αυξάνονται τα έσοδα του κράτους βάσει ενός φόρου παράνομου. Και επαναλαμβάνω, δεν τηρείται καν η αρχή της αναλογικότητας. Και εδώ επικαλούμαστε την συνθήκη της Ρώμης που αναφέρει ότι θα πρέπει οι τελεωνιακοί δεσμοί και οι αντίστοιχοι φόροι να εξαλειφθούν. Τι έγινε εδώ, τίποτα από αυτά δεν εφαρμόστηκε και ουσιαστικά βρήκαν έναν τρόπο να επιβάλλουν ένα φόρο στους πολίτες ε, και τα ποσά αυτά να πάνε στα ταμεία του κράτους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από όσα άκουσα, ε, καλό θα ήταν να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Η Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να δει τι άλλο μπορεί να κάνει. Υπάρχει διαδικασία επιπαραβάση που συνεχίζεται αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν, δεν αφορά ακριβώς αυτό το ζήτημα, όπως είπε και η Επιτροπή. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω πληροφορίες από την Κομισιόν από αυτού και εφόσον πρόκειται για τόσο ευαίσθητο ζήτημα, αλλά και ότι είναι επίγον να δοθούν απαντήσεις, θεωρώ ότι ο συντονιστή θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω το θέμα και να δούμε έτσι πώς θα μπορέσει η Επιτροπή μας να δώσει μια δημόσια απάντηση. Ο συντονιστή όμως θα πρέπει να το κοιτάξει πρώτα αυτό. Και θα πρέπει εκείνος να πάρει μια απόφαση. Γιάννη. Βεβαίως. Οι αναφέροντες όμως δεν πρέπει να γυρίσουν στην πατρίδα τους με την εντύπωση ότι δεν γίνεται τίποτα και εμείς θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη κατάσταση και εμείς πρέπει να συντάξουμε επιστολή προς τις Ιρλανδικές αρχές και θα με ενδιέφερε να δω πώς αιτιολογούν αυτά που κάνουν εκεί. Συμφωνώ κατά τα άλλα με την ε, πρότασή σας ε, να δημοσιοποιήσουμε την προβληματική αυτή και να συζητήσουμε και με προφορική επερώτηση το θέμα στο Κοινοβούλιο. Εντάξει. Συμφωνείτε να συζητηθεί στη συνάντηση των ε, συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ τους αναφέροντες. Τελειώσαμε με το σημείο αυτό και προτείνω να περάσουμε στο επόμενο. Είναι το σημείο 18. Πρόκειται για την 1211 του 2009 αναφορά που έχει υποβληθεί από τον Λέον Μπρέτο και την 1053 του 2010 Αντώνιο Σουζάνα Βιβέλη Πρόκειται για θέματα διπλής φορολόγησης στην Ιταλία και στη Γερμανία. Και μια απόφαση που αφορά τη Γερμανία και τη Γαλλία. Οι αναφέροντες της δεύτερης αναφοράς έχουν το λόγο ο κύριος Αντώνιο Κιφέλη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Αντώνιο Κιφέλη και εδώ και 42 χρόνια μένω στη Γερμανία. Εδώ και 33 χρόνια οδηγώ το όχημά μου και μεταφέρω εμπορεύματα στην Ιταλία. Εδώ και πολλά χρόνια είμαι φορολογούμενος δίπλα και στις δύο χώρες και πρέπει να σας πω ότι ο εργοδότης μου πληρώνει εισφορές στην Ιταλία, αρνούμε όμως σήμερα αυτήν την διπλή φορολόγηση. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορώ πλέον να ανταποκριθώ. Η γυναίκα μου εργάζεται στη Γερμανία και ένα τμήμα του μισθού της ε, έχει κατασχεθεί. Έχω επίσης χάσει το όχημά μου, ένα εμπορικό όχημα και τελικά πληρώνω 350, 350 ευρώ το μήνα στην ε, στις γερμανικές φορολογικές αρχές. Μετά από πολλές δαπάνες και πολλές έρευνες, οι Ιταλικές φορολογικές αρχές μου απάντησαν ότι ο εργοδότης μου είναι Ιταλός, πληρώνει τις εισφορές του στην Ιταλία, δεν μπορούν λοιπόν να μου επιστρέψουν ε, τη φορολογία. Έχω καταστραφεί οικονομικά και εγώ και η γυναίκα μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ από πλευρά Επιτροπή. Μαρίνα Whitehouse. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον αναφέροντα για την παρουσίασή του. Πολύ σύντομα θα ήθελα να παρουσιάσω την δική μας ε, ε, προσέγγιση. Ο αναφέρον είναι Ιταλός πολίτης, αλλά διαμένει στη Γερμανία. Τα, και, τα ζωτικά του συμφέροντα, θέλετε, βρίσκονται στη Γερμανία. Ως εκ τούτου είναι Γερμανός προλογούμενος έτσι, η Γερμανία έχει το δικαίωμα να φορολογήσει το εισόδημά του. Ο αναφέρον κύριος Τσιφέλη είναι ε, οδηγός φορτηγού μακρινών αποστάσεων και έτσι ασκεί τις δραστηριότητε του όχι μόνο στη Γερμανία, ούτε μόνο στην Ιταλία, αλλά στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάνω από έξι μήνες το χρόνο ε, ταξιδεύει μεταξύ Γερμανίας, ε, Ισπανίας, Γαλλίας, αλλά όχι στην Ιταλία και τα Σαββατοκύριακα τα στη Γερμανία με την οικογένειά του. Το γεγονό ότι ο κύριο Τσιφέλη ε, είναι υπάλληλο μια Ιταλική ε, εταιρεία θεωρείται αρκετό στοιχείο για την Ιταλική κυβέρνηση για να ε, φορολογήσει το 100% του εισοδήματός του. Ωστόσο, η Γερμανία επίσης τον φορολογεί γιατί διαμένει στη Γερμανία. Το φορολόγει λοιπόν επ' αυτού του εισοδήματο χωρίς καμία ε, έκπτωση φόρου. Ο αναφέρον έχει ζητήσει αποζημίωση από τις ταλικές αρχές, αλλά δεν του έχει χορηγηθεί. Και οι γερμανικές αρχέ, οι ε, φορολογικές αρχές έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία ε, συμφωνίας, αμοιβαία συμφωνίας. Τι συμβαίνει λοιπόν εάν ένα κράτο μέλο ε, είναι υπάλληλο σε, ε, σε ένα κράτο μέλο, αλλά ασκεί τι δραστηριότητέ του σε ένα άλλο κράτο μέλο. Συνήθω τα κράτη-μέλη έχουν συνάψει ε, συμφωνίε διπλή φορολόγηση όπου κατανέμουν τα, τα δικαιώματα φορολόγησή του. Έτσι έχουν καταλήξει μεταξύ του σε μια συμφωνία για το πώ θα φορολογήσουν ε, τους πολίτες που ε, ε, έχουν δραστηριότητε και στις δύο χώρες. Υπάρχει μια τέτοια συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας. Στο άρθρο 15 για τις εξαρτημένες υπηρεσίες κατανέμονται τα δικαιώματα φορολόγησης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διπλή φορολόγηση στην οποία επόκειται ο φορολογούμενος οφείλεται απλά και μόνο στην ερμηνεία ε, το, της Γερμανίας και της Ιταλίας των διατάξεων αυτή τη σύμβαση. Δεν υπάρχει κάποια διάταξη στη συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκής Ένωση που να δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα να αναλάβει δράση εδώ και δεν υπάρχει κάποια διάταξη για την εξάλληψη της διπλής φορολόγησης. Δυστυχώς λοιπόν αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ε, ότι η διπλή φορολόγηση αποτελεί εμπόδιο στην εσωτερική αγορά, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Ε, Ευχαριστώ. Θα πέσουμε τον κύριο Ροκατάγια. Πριν όμως σας δώσω το λόγο, Υπάρχουν και άλλες αναφορές, τέσσερις στο σύνολό τους, που αφορούν το ίδιο θέμα, την διπλή φορολόγηση. Η τέταρτη αφορά μια σύγκρουση μεταξύ Γερμανίας και Πορτογαλίας. Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ αναφέρομαι στην υπόθεση Μπρεύτο που δεν είναι ίδιο με την υπόθεση Τσιφέλη. Βάσει των τελευταίων ε, πληροφοριών ε, που έχει υποβάλει ο υπογράφων την αναφορά στο κοινοβούλιο, δεν πρόκειται για διπλή φορολόγηση. Ο αναφέρον θεωρεί ότι πρόκειται για διάκριση διακριτική μεταχείριση. Και πρόκειται εδώ για μία διμερή συμφωνία, για να επαναλάβω κάτι που ίδια, ήδη ακούσαμε στην αίθουσα, πρόκειται για άμεση φορολογία και σαφώς θα αναφέρω και εγώ την αρχή της επικουρικότητας, την αρχή της αναλογικότητας. Πρόκειται για αρμοδιότητες των κρατών μελών και η φορολογία, όπως ξέρετε, έχει εναρμονιστεί σε ένα πολύ περιορισμένο τμήμα της και για να αλλάξει η κατάσταση αυτή θα πρέπει να υπάρξει ομοφωνία των κρατών μελών. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί το θέμα της φορολογίας είναι εξαιρετικά ε, ευαίσθητο, εξαιρετικά λεπτό για όλα τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα σήμερα εν ώψη της οικονομικής κρίσης. Η υπόθεση Μπρεύδο λοιπόν ουσιαστικά ε, πρόκειται για έναν Γερμανό υπήκο, ο οποίος ζει στη Γερμανία, εργάζεται όμως στο γαλλικό δημόσιο τομέα. Ένας πραγματικό Ευρωπαίος πολίτης, αν θέλετε. Το 1959 η διμερή σύμβαση μεταξύ της Γερμανίας και της Γαλλίας προβλέπει ότι άτομα διαφορετικής εθνικότητας που εργάζονται για το δημόσιο τομέα της άλλης χώρας, τότε υπήρχαν ελάχιστα άτομα, κυρίως ε, διπλωμάτες αφορούσε αυτή η διμερή σύμβαση. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις ε, των ατόμων αυτών που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι έχοντας διαφορετική υπηκότητα από τη χώρα στην οποία εργαζόταν. Η φορολόγηση λοιπόν στη Γερμανία θα ήταν μεγαλύτερη από αυτή που επιβάλλεται στη Γαλλία. Ένας συνάδελφος ε, ο οποίος θα εργαζόταν αντιστοίχως στο γαλλικό δημόσιο τομέα θα πλήρωνε 50% αυτών που πληρώνει ε, ο αναφέρον στη Γερμανία. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι σαφής όμως για τέτοιες υποθέσεις. Διαφορετική φορολόγηση στα διαφορετικά κράτη-μέλη και η διμερή σύμβαση εδώ διέπει τα θέματα των ε, ατόμων που εργάζονται στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα. Γίνεται επίσης διάκριση μεταξύ των διασυνοριακών περιοχών και των υπολείπων περιοχών Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορεί να θεωρηθούν διακριτική μεταχείριση. Υπάρχει επίσης και η υπόθεση Τσίλη του 1978, η οποία είναι παρόμοια με την... η οποία, συγγνώμη, είναι διαφορετική με την σημερινή υπόθεση. Ο κύριος Μπρεύντο, όπως αναφέρει ο ίδιος, δεν είναι αντικείμενο διπλής φορολόγησης, δεν υπάρχει επίσης διακριτική μεταχείριση, καθότι τα κράτη-μέλη έχουν αποφασίσει σε μια διμερή σύμβαση την χρησιμοποίηση του κριτηρίου της υπηκότητας έτσι ώστε να κατανείμουν τις αρμοδιότητες σε θέματα φορολόγησης. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θεωρεί ότι η κατανομή αυτή των φορολογικών αρμοδιοτήτων είναι ορθή. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Φιλίπς Βίταλα για την αναφορά Γκέρχαρτ Χάινς. Ναι, ευχαριστώ. Η αναφορά του Γκέρχαρτ Χάινς αφορά την αμοιβαία αναγνώριση εγγράφων από τις αρχές των κρατών μελών. Ο αναφέρον ισχυρίζεται ότι οι γερμανικές φορολογικές αρχές δεν αναγνωρίζουν τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι η σύζυγός του δεν είχε εισοδήματα στην Πορτογαλία και φαίνεται ότι δεν αναγνωρίζουν το έγγραφο που εξέδωσαν οι πορτογαλικές αρχές. Από την άλλη πλευρά, οι πορτογαλικές αρχές φαίνεται να μην αναγνωρίζουν το έγγραφο που εξέδωσαν οι γερμανικές φορολογικές αρχές. Και το θέμα αυτό δεν αφορά τη διπλή φορολόγηση, αλλά μάλλον για ε, ε, την καλή συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών δύο κρατών μελών. Η υπόθεση μπορεί να εξεταστεί και μέσα από το πρίσμα της οδηγίας αμοιβαίας αρρωγής, η οποία υπάρχει και στα πλαίσια της οποίας οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών θα έπρεπε και μπορούν να συνεργάζονται για να αποφεύγουν την ε, διπλή μη φορολόγηση των ε, Ευρωπαίων φορολογουμένων. Ένα άλλο θέμα είναι ότι οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα με την εφαρμογή των συμβάσεων για τη διπλή φορολόγηση. Το θέμα όμως αυτό είναι της εθνικής αρμοδιότητας των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Αυτό που μπορούμε να συμβουλεύσουμε εδώ, τον φορολογούμενο, τον αναφέροντα εν προκειμένου, είναι να ζητήσει τη βοήθεια από την Solvit που είναι μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βοηθάει σε περιπτώσεις προβλημάτων συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών. Όπως είπε ο συνάδελφος, η διπλή φορολόγηση θεωρείται ως πρόβλημα εσωτερικής αγοράς από την Κομισιόν. Η Κομισιόν όμως η ιδία δεν έχει εξουσία να χειριστεί το θέμα της διπλής φορολόγησης ε, έτσι όπως έχει τώρα το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να ακούσουμε και για την υπόθεση Άξελ Έγκαιμαν να πιάσουμε και τα τέσσερα. Στην περίπτωση Άξελ Έγκεμαν πρόκειται περί Γερμανού υπηκόου ο οποίος για κάποιο διάστημα ε, παρέμεινε στη Γαλλία, ε, ήταν σε κάποια υπηρεσία υγείας, σε κάποιο Ινστιτούτο Υγείας, έμεινε εκεί, μετά αποφάσισε να ξαναγυρίσει πίσω στη Γερμανία και να εργαστεί. ως ε, ανεξάρτητος, όχι ως μισθωτός και φορολογήθηκε στη Γερμανία. Δεν υπάρχουν όλες οι πληροφορίες στην αναφορά, νομίζω, αλλά η Γερμανία θεώρησε ότι αφού ήταν κάτοικος διέμενε στη Γερμανία θα έπρεπε να φορολογεί εκεί. Η Γαλλία όμως συνέχισε να τον φορολογεί και ο μόνος τρόπος που βρήκε για να λύσει το πρόβλημά του ήταν να ξαναπάει στη Γερμανία, να εγκατασταθεί εκεί, επίσης για να αποφύγει τη, τη διπλή φορολόγηση. Η Κομισιόν κατανοεί την ε, κατάσταση, το πρόβλημα. Θεωρούμε ότι η διπλή φορολόγηση είναι πολύ βλαβερό πράγμα στην ε, ενιαία αγορά αλλά και εδώ πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη με τις φιλικές διαδικασίες που προβλέπουν οι διμερείς συμβάσεις πρέπει να βρουν μια λύση. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι είναι υπόθεση των κρατών μελών. Εκείνα θα πρέπει να λύσουν αυτά τα προβλήματα διπλής φορολόγησης και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν διμερείς συμβάσεις για αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βουλάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να απαντήσω σφαιρικά χωρίς να αναφερθώ στις συγκεκριμένες αναφορές παρόλο που έχουν ορισμένα κοινά σημεία σχετικά με την ε, διπλή φορολόγηση. Πράγματι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η διπλή φορολόγηση ε, αφορά τις ε, συμβάσεις που έχουν ε, υπογραφεί μεταξύ των κρατών μελών και ενδεχομένως όπως υπόθηκε και από την Επιτροπή υπάρχει δυνατότητα φιλικής επίλυσης ε, των προβλημάτων αυτών και σίγουρα και αναφέροντες έχουν κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς να έχουν επιτύχει κάποιο αποτέλεσμα, γι' αυτό και έχουν έρθει ενώπιον μα σήμερα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι πράγματι αυτή η σύμβαση για την διπλή φορολόγηση, η συμφωνία διπλής φορολόγησης, είναι δίκαιη και αν τα, οι καταγγελίες και τα, τα παράπονα του αναφέρονται μπορούν να γίνουν παραδεκτά. Πράγματι, εκτός από την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας, ξέρουμε ότι αυτή η διπλή φορολόγηση πλήττει ε, την ε, ενιαία αγορά. Τώρα, όπως είπε και η Επιτροπή, καθώς η Επιτροπή είπε ότι δεν έχει αρμοδιότητες επί του θέματος, Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ένα-δύο άρθρα τη Συνθήκη Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 46α και β σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων ανθρώπων ε, και υπηρεσιών, ε, διασφαλίζει την στενή συνεργασία μεταξύ των ε, εθνικών αρχών για την κατάργηση των κακών πρακτικών ε, με στόχο την απελευθέρωση της κυκλοφορίας και κίνησης ε, των ε, ατόμων και των εργαζομένων. Στο 49 λοιπόν, εάν την πληροφορολόγηση απαγορεύεται λοιπόν. Στο άρθρο 50 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ασκούν τις δραστηριότητε και τις αρμοδιότητες που τους έχουν χορηγηθεί διασφαλίζοντας την συνεργασία σε επίπεδο εθνικής διαχείρισης ε, και, και, και, και καταργώντας ε, αυτές τις κακές πρακτικές που ε, παρατηρούνται, που παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η Επιτροπή εδώ θα πρέπει να ε, εντοπίσει τις ανισότητες ε, που δημιουργούνται εδώ. Και εφόσον δεν υπάρχει ένα μήνυμο, ένα ελάχιστο ε, κοινωνικών και δημοσιονομικών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών και σχετικά με αυτή την διπλή φορολόγηση μπορούμε να προτείνουμε να υπάρχει μία φορολόγηση στον, ε, στη χώρα διαμονής του εργαζομένου, φορολόγηση επί, και μια φορολόγηση επί του εισοδήματος στον χώρο εργασίας του εργαζομένου. Την στην πρώτη περίπτωση, για παράδειγμα, ο αναφέρον είναι ε, οδηγός φορτηγού. Ε, το γεγονός ότι εργάζεται σε πολλές χώρες τι σημαίνει, πού θα πρέπει να τον ε, φορολογήσουμε. Και αυτή η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί για όλους ε, ε, τους εργαζομένους που αλλού εργάζονται και αλλού διαμένουν. Υπάρχει λοιπόν μια συμβατότητα εδώ. Και μια λήψη συνοχής μάλλον και για την ε, φορολόγηση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθείτε η ε, η επαγγελματική έδρα του υπαλλήλου χωρίς αυτό να ε, σημαίνει ότι δεν μπορεί να φορολογηθεί και στην χώρα διαμονής του. Αυτό απλώς να μην υπάρχει μια σώρευση για τον δύο. Θα πρέπει λοιπόν να αποστέλουμε μια επιστολή στις αρμόδιες αρχές για να ικανοποιήσουμε το αίτημα του αναφέροντα. Ευχαριστώ για Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Μπελόν Θέλουμε ελεύθερη κυκλοφορία, εσωτερική αγορά, κυκλοφορία αγαθών, κεφαλαίων και προσώπων. Και εδώ βλέπουμε τα κράτη-μέλη να δημιουργούν νέα σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει μόνο την, το δικαίωμα, αλλά την υποχρέωση να επιληθεί του θέματος ένα κράτος μέλος εδώ, στο οποίο διαμένει κάποιος, εργάζεται όμως σε μια άλλη χώρα και η έδρα της εταιρεία στην οποία εργάζονται βρίσκεται σε μια τρίτη χώρα, αυτό πλέον θα γίνει καθημερινότητα. Αυτό σημαίνει ελεύθερη κυκλοφορία. Και βεβαίως αυτό πρέπει να αλλάξει εδώ είναι το δίκαιο που αφορά τη φορολογία. Όλα τα κράτη-μέλη βεβαίως έχουν διαφορετική φορολογία και σήμερα εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο σήμερα να γίνει αυτό. Αλλά το πρώτο βήμα θα ήταν να επιβληθεί ένα κοινότικό φόρο, αλλά αυτό που ήδη σήμερα έχουμε πληρώσει θα πρέπει να συνυπολογίσει. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε δύο φορέ. Και εάν εγώ παραδείγματο χάρη εργάζομαι σε μια χώρα και μένω στη Γερμανία, δεν μπορώ να ξαναπληρώνω φόρο στη Γερμανία να έχω πληρώσει ήδη για την επαγγελματική μου δραστηριότητα εκεί όπου εργάζομαι. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εσωτερική αγορά θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ενιαία κατάσταση όσον αφορά τη φορολογία. Η κατάσταση είναι παράλογη σήμερα, η διπλή φορολογία είναι παράδεκτη. Και πρόκειται για θέμα ερμηνείας. Αυτό που λένε σήμερα τα κράτη-μέλη είναι ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μπορούμε. Αλλά αυτό δεν γίνεται εις βάρος των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Δηλαδή τελικά δεν συμφωνούν τα κράτη-μέλη και επιβάλλονται διπλή φορολογία στα κράτη, στους Ευρωπαίους πολίτες από τα κράτη. Τώρα το θέμα της φοροδιαφυγής, τα ποσά είναι τεράστια. Αυτό όμως είναι κάτι άλλο. Όσο δεν συμφωνούν πάντως τα κράτη-μέλη για τα θέματα αυτά και δεν υπάρχει ενιαία φορολόγηση, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Επαναλαμβάνω, η Επιτροπή δεν έχει απλώς το δικαίωμα, αλλά την υποχρέωση να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Άκουσα την πρόταση να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και αναφέρθηκε επίσης και το Solvit. Πρέπει να το κάνουμε, δεν πρέπει. Δεν πρέπει όμως να επιβάλλουμε στον αναφέροντα να ξαναρχίσει τη διαδικασία από την αρχή. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει ίσως οι αναφέροντες οι οποίοι έχουν υποβάλει την αναφορά τους να βρουν μια λύση από μας. Δεν μπορεί σήμερα ένας φορολογούμενος να του επιβάλλεται 65% των εισοδημάτων του να φεύγουν σε φορολογία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ίσως ε, αυτό θα μας οδηγήσει σε μια ενιαία λύση, σε μια συμβαστική λύση. Τελειώνοντας λοιπόν θέλω να σας πω ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια αδυναμία η εσωτερική αγορά δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και θα πρέπει να βρούμε λύση για όλα αυτά τα φορολογικά προβλήματα. Τελειώς δεν λειτουργεί η εσωτερική αγορά. Τι μπορούν να κάνουν σήμερα οι αναφέροντες οι οποίοι μένουν κάπου, εργάζονται κάπου αλλού. Νομίζω ότι αυτό που ουσιαστικά θα αποτελέσει και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί σήμερα λόγω φορολογικών θεμάτων να εμποδίζεται. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω αναφέρον. Μικρόφωνο, μίνουτο. Ένα πράγμα θα ήθελα να πω μόνο. Νιώθω ότι διχάνω διακριτική μεταχείριση από τι ε, γερμανικέ φορολογικέ αρχέ. Γιατί οι συνάδελφοί μου που εργάζονται στη Γερμανία δεν φορολογούνται. Και αυτό εμένα ε, με προβληματίζει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ αυτών των αναφορών αλλά και διαφορές. Γι' αυτό και θα πρέπει να συνεχίσουμε την εξέτασή τους και όπως ε, ε, πρότεινε και ο κύριος Γιάς. Θα μπορούσαμε να καλέσουμε τις εθνικές ε, αρχές, τις αρμόδιες εθνικές αρχές, Να τις καλέσουμε εδώ λοιπόν στην Επιτροπή μας ε, για να μπορέσουμε να τους ε, μιλήσουμε για τα προβλήματα αυτά. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Αφήνουμε λοιπόν ανοιχτές τις ε, αναφορές και θα, θα, ρωτήσουμε, θα ζητήσουμε μάλλον από τις εθνικές αρχές να έρθουν εδώ. Ευχαριστούμε, ας προχωρήσουμε. Αυτό είναι σημαντικό για τους αναφέροντες μπορούμε και εμείς ως Επιτροπή ε, να παρέμβουμε. Δεν ξέρω διαδικαστικά ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα, θα προσθέσουμε μία κοινοποίηση στην Solvit και θα τους ρωτήσουμε να κάνουν ό,τι μπορούν. David. Αυτό που κάνει η Solvit είναι να διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο κρατών μελών. Αν υπάρχει επικοινωνία είναι περιττό να παρέμβει και το Solvit θα έλεγα. Επίσης ε, νομίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία με την Κομισιόν όταν υποβάλλουμε αναφορές για να τις εξετάσουν. Δεν θα έρχονται λίγους μήνες μετά την υποβολή και θα, να μας λένε να πάμε στην Solvit. Η Solvit είναι της Κομισιόν και αν πιστεύουν ότι είναι εναλλακτική αυτή μπορούν να το προβλέψουν εκείνοι. Δεν είναι δική μας δουλειά να πούμε στους αναφέροντες «Α, συγγνώμη, καλύτερα να πάτε στο Solvit». Αυτό το στάδιο το έχουμε ξεπεράσει. Ο κύριος Μπουλάν. Η πρόταση να ε, καλέσουμε τα κράτη-μέλη μου φαίνεται ε, σωστή, ωστόσο δεν πρέπει να σταματήσουμε σε αυτές τις τέσσερις αναφορές και να μείνουμε σε αυτές, θα πρέπει να ε, έρθουμε σε επαφή με, ε, με όλα αυτά τα κράτη-μέλη που εμπλέκονται σε διαδικασίες διπλής φορολόγησης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ε, Ευχαριστώ. Θα στείλουμε ένα γραπτό αίτημα, μια γραπτή πρόσκληση και ελπίζουμε να λάβουμε και γραπτή απάντηση. Σε ό,τι αφορά τη Solvit, νομίζω ότι ο David έχει δίκιο. Όπως και να έχει όμως μπορούμε να στείλουμε μια επιστολή στην ε, Solvit, επισημένοντας ε, τα ζητήματα αυτά και ζητώντα του να δουν τι μπορούν να κάνουν. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, Μπορούμε να το κλείσουμε αυτό το ζήτημα. Α, η Επιτροπή. Πολύ σύντομα. Ήθελα να απαντήσω στις προτάσεις του κυρίου Γιάου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει καταβάλει προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα. Γνωρίζουμε ότι το να έχουμε 27 κρατημέλη και 27 διαφορετικά φορολογικά συστήματα οδηγεί σε ε, επικαλύψεις που μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιες συγκεκριμένες υποθέσεις διπλής φορολόγησης που συχνά φτάνουν μέχρι την Επιτροπή Αναφορών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, ε, όπως αναφέρει ο κ. Τσιβέλη, όπου δεν υπάρχει φορολόγηση. Αλλά βεβαίως και δεν, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε η Επιτροπή Αναφορών ακούει ποτέ τίποτα, κανένα παράπονο για αυτές τις ε, υποθέσεις. Αυτή η κατάσταση όμως οφείλεται στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ε, προτείνει μια ανακοίνωση τον τελευταίο Δεκέμβριο για τα εμπόδια που τίθενται στην ε, διασυνοριακή ε, δραστηριότητα αναφερόμασταν και στην διπλή φορολόγηση εκδώσουμε και ανακοίνωση τον Ιούλιο, συγκεκριμένα για το, αυτό το θέμα της διπλής φορολόγησης και για του χρόνου πιθανόν προγραμματίζουμε να ε, υποβάλουμε μια συγκεκριμένη πρόταση που θα εστιάζει σε ένα μηχανισμό που θα απαχρεώνει τα κράτη-μέλη ε, στην εξέβρεση φιλικών διαδικασιών για την εξέβρεση μιας λύσης δεν μα ενδιαφέρει ποια θα είναι αυτή η λύση, αρκεί να υπάρχει μια λύση στο ζήτημα της διπλής φορολόγηση. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, για τις πληροφορίες. Ας ε, προχωρήσουμε στο σημείο 19. Ε, αναφορά του Pierre Gerard, Βελγική Εθαγένεια, εξ ονόματο της Επιτροπής για την Υπεράσπιση των Βέλγων Μεθοριακών Εργαζομένων που εργάζονται στη Γαλλία, σχετικά με τη φορολόγηση των γαλλικών συμπληρωματικών συντάξεων στο Βέλγιο και μετά ε, αναφορά του Αρσέν Σμιτ ε, σχετικά με τη φορολόγηση στη Γερμανία των ε, συντάξεων συνταξιούχων και συνοριακών εργαζομένων που διαμένουν στη Γαλλία. Ο Πιάρ Ζεγάρ είναι εδώ, του δίνω το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Λέγομαι Πιέρ Ζεγάρ και καταρχήν θα ήθελα να σας δώσω κάποια συμπληρωματικά στοιχεία για να σας παρουσιάσω την υπόθεση αυτή που έχουν υποβάλει η Ένωση, της οποίας είμαι πρόεδρος, των διασυνοριακών εργαζομένων, η οποία υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στο Βέλγιο. Όσον αφορά τους συνταξιούχους και μέλλοντες συνταξιούχους οι οποίοι διαμένουν στο Βέλγιο, οι οποίοι όμως εργάστηκαν ή εργάζονται στην ε, Γαλλία, θα πρέπει να εξετάσουν τη σημερινή φορολόγηση των επικουρικών συντάξεων ατόμων που διαμένουν στο Βέλγιο αλλά έχουν εργαστεί στην Γαλλία. Θα ήθελα λοιπόν να προσελκύσω την προσοχή σας τα εξής. Πρώτον, πέρασαν 40 χρόνια μέχρι να υπάρξει μια αναθεώρηση της σύμβασης του 64 μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου, κάτι που ζητούσαμε διαρκώς στην Ένωσή μας, για τα άτομα αυτά που φορολογούνται στο Βέλγιο για μια επαγγελματική δραστηριότητα στη Γαλλία. Αποτέλεσμα αυτής της αναθεώρησης, σημερινή σύνταξη, όχι τους οποίους εκπροσωπούμε, πλήρωσαν φορολογία εισοδήματος στο Βέλγιο παρανόμως, καθότι διαμένουν σε μια χώρα η οποία δεν αναθεώρησε αυτήν την σύμβαση που υπάρχει από το 1964 και δεν θα επιμείνω περισσότερα στα ποσά, στα δισεκατομμύρια που απέφερε αυτή η δραστηριότητα στην οποία διαμένουμε. Δυστυχώς δεν μπόρεσε αυτή η νέα ε, αναθεώρηση της φορολογίας να επιβληθεί στους νέους συνταξιούχους. Υπάρχει λοιπόν σήμερα ένα status quo το οποίο, στο οποίο βασίζεται η σημερινή μας αναφορά. Τρίτον, οι συνέπειες για τους συνταξιούχους είναι πολύ σοβαρές και ελπίζαμε σαν ε, αντιστάθμισμα η φορολογία των επικουρικών συντάξεων της Γαλλίας από το βελγικό κράτος τουλάχιστον να ανταποκρίνονται στις διατάξεις ε, της φορολόγησης των συντάξεων βάσει του δεύτερου πυλώνα, όμως από την 1η Ιανουαρίου του 2004 βάσει του βελγικού νόμου και της δημοσίευσής τους του 2009 οι βελγικές φορολογικές αρχές θα μπορούσαν να είχαν μειώσει σημαντικά τη φορολόγηση των συντάξεων κάτι το οποίο δεν γίνεται ιδιαίτερα όσον αφορά τις επικουρικές συμβάσεις από το βελγικό κράτος σε εργαζόμενους στη Γαλλία αλλά και σε άλλα γειτονικά κράτη. Ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να αλλάξει τη στάση του βουλικού κράτους για το θέμα αυτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ και επαναλαμβάνω μια τελευταία φορά. Πραγματικά οι διασυνοριακοί συνταξιούχοι και εργαζόμενοι ελπίζουν στην ε, παρέμβασή σας η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ τον αναφέροντα. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για ένα θέμα φορολόγησης στη χώρα διαμονής βάσει του βελγικού νόμου ενισχύει φορολογούνται οι συντάξεις στη χώρα διαμονής του συνταξιούχου. Αυτό εξάλλου παρουσιάστηκε και στην πρώτη απάντηση της Επιτροπής τον Ιανουάριο, όπου διατυπώνουμε ότι τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για να καθορίσουν είτε μονομερός είτε με διμερείς συμβάσεις την φορολογική Πολιτικοί που θα ακολουθήσουν. Σήμερα το κοινοτικό δίκαιο δεν εμποδίζει την φορολόγηση στο Βέλγιο γαλλικών συντάξεων. Όσον αφορά το δεύτερο σημείο, φορολόγηση στο Βέλγιο των επικουρικών συντάξεων από γαλλικά ταμεία, σύμφωνα με την φορολογία που ισχύει στο Βέλγιο για τις βελγικές επικουρικές συντάξεις. Ακούσαμε ότι υπήρξε αναθεώρηση του βελγικού νόμου που αφορά τη φορολόγηση των επικουρικών συντάξεων. Η Γενική Διεύθυνση Ταξούντ, η οποία βεβαίως έχει και τη σύμφωνη γνώμη της νομικής υπηρεσίας της Επιτροπής, θεωρεί ότι αυτές οι αλλαγές αφορούν κάποια μεταβατικά μέτρα όσον αφορά την αναθεώρηση, μετά δηλαδή την πληροφορία του νόμου του 2003. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό και θα σας παρουσιάσω τώρα το σημερινό, το ισχύον σύστημα φορολόγησης και θα δω κατά πόσο αυτό είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο. Στο βελγικό νόμο για τη φορολόγηση των συντάξεων δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ επικουρικών συντάξεων βελγικών και άλλων. 10% είναι η φορολόγηση για τις εργοδοτικές εισφορές στο κεφάλαιο βάσει του συστήματος της κεφαλαιοποίησης και 70% και 16% φορολόγηση όσον αφορά τις εισφορές των εργαζομένων. Η απόδοση της τάξης του 3% επίσης φορολογείται όταν πρόκειται για επενδύσεις σε ακίνητα. Η φορολόγηση τώρα των ε, γαλλικών συντάξεων γίνεται με διαφορετικό τρόπο καθότι υπάρχει μια διαφορετική, αν θέλετε, διαφορετικός σχεδιασμός του συνταξιοδοτικού συστήματος στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Τι εννοώ. Το Βέλγιο οργανώνει το σύστημα φορολόγησης σε τρεις πυλώνες. Ο δεύτερος πυλώνας που αφορά τις επικουρικές συντάξεις προέρχεται από ένα σύστημα που βασίζεται στην κεφαλαιοποίηση. Δεν είναι λοιπόν υποχρεωτικό ούτε για τις επιχειρήσεις. Απλώς μπορεί να προτείνει στους εργαζόμενους μία συμμετοχή στο σύστημα αυτό που απορρέει από το δεύτερο πυλώνα. Ενώ αντίθετα τα συστήματα επικουρικής ε, σύνταξης στην Γαλλία ανταποκρίνονται πολύ περισσότερο στην πρώτο πυλώνα. Πρόκειται δηλαδή για μία φορολόγηση σταδιακή. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συμπληρωματικές, οι επικουρικές συντάξεις είναι τελείως διαφορετικές στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορετική μεταχείριση του βελγικού νόμου και θεωρούμε ότι εδώ δεν υπάρχει παραβίαση του κοινοτικού νόμου και φορολογούνται στο Βέλγιο οι γαλλικές συντάξεις με διαφορετικό τρόπο βάσει της σύμβασης που έχει υπογραφεί διμερός από την Γαλλία και το Βέλγιο για θέματα φορολογίας και αυτό οφείλεται στο ότι τα δύο συστήματα είναι διαφορετικά στο Βέλγιο και στη Γαλλία έτσι και αλλιώς πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Θα ήθελε κάποιος να πάρει το λόγο. Όχι. Θα δώσω το λόγο στον αναφέροντα, αλλά σύντομα μπορείτε. το πρόβλημα παραμένει το ίδιο και η λύση παραμένει η ίδια. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι συνταξιούχοι μεθοριακοί εργαζόμενοι καθ' όλη τη διάρκεια της ε, καριέρας του, της ε, επαγγελματικής του ε, πλήρωναν φόρου στο Βέλγιο. Ε, και έτσι τώρα έχουμε μια διαφορετική κατανομή των συντάξεων, αλλά εμείς ε, στο Βέλγιο δεν έχουμε καμία ε, σύνταξη, μόνο τη γαλλική σύνταξη λαμβάνουμε, η οποία μας ε, ε, δίδεται υποχρεωτικά. Ένα, κατά μέρος λοιπόν από τον εργοδότη, από, κατά ένα άλλο μέρος από τους υπαλλήλους σε άλλε χώρε όπου οι κάτω χώρες, στο Λουξεμβούργο και στη Γερμανία, εκεί ο συνταξιούχο πληρώνει φόρου ε, στην χώρα που εργαζόταν. Στη Γαλλία, ο υπάλληλο πληρώνει φόρου ε, στη Γαλλία και ο συνταξιούχο στο Βέλγιο. Τέλος, είπα ότι δεν υπάρχει μια είναι αφήσει και αυτή η σύνδεση γιατί απαιτείται ένα ελάχιστο, δηλαδή η γαλλική επικουρική σύνταξη θα πρέπει να αλλάξει και να, να γίνει σαν την βελγική επικουρική σύνταξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουν τεθεί πολλά ζητήματα σε ό,τι αφορά την αρχή της επικουρικότητας και αρμοδιότητας των κρατών μελών. Ωστόσο, ακόμα και η απάντηση της Επιτροπής ε, επιβεβαιώνει την ύπαρξη προβλήματος. Η Επιτροπή λέει ότι πρόκειται για πρόβλημα εθνικής δικαιοδοσίας, όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να αποστείλουμε ένα σημείο μας στις εθνικές αρχές, εξηγώντας ε, το ζήτημα. και να τους ζητήσουμε να προσπαθήσουν να επιλύσουν ε, τα προβλήματα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ως Επιτροπή Αναφορών. Θα γράψουμε λοιπόν, ε, αποστείλουμε ένα αίτημα προς τις Εθνικές Αρχές. Ευχαριστούμε πολύ. Προχωρούμε στο ε, σημείο 22 αιτήσεις, άρα αναφορές συγγνώμη έχουμε εδώ, παρόμοιες. Η πρώτη για να φέρουσα είναι παρούσα. Κυρία Χενρίκα Μαγδαλένα Άντερσεν. Έχει το λόγο. Αλλά θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι, γιατί έχουμε ακόμα τρεις αναφορές στην μεσηγεία μας διάταξη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω όλους. Δεν μπορώ να συνοψίσω βέβαια το περιεχόμενο της αναφοράς σε πέντε λεπτά. Δύο αναφορές πρέπει να υποβάλω για διακριτική μεταχείριση από τις δανεικές αρχές προς άλλους πολίτες και άλλων χωρών που διαμένουν στη Δανία. Πρόκειται για ανθρώπους που παίρνουν σύνταξη επίδομα αναπηρίας και αυτό το επίδομα υπολογίζεται με τρόπο διαφορετικό από ό,τι οι συντάξεις που καταβάλλονται σε πρόσωπα που δεν έφυγαν ποτέ από τη Δανία για να εργαστούν αλλού. Το θέμα έχει ως εξή τώρα. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί μέθοδοι υπολογισμού. Για το συγκεκριμένο επίδομα υπάρχουν οι δανείοι υπήκοοι που παίρνουν ένα ποσό από αυτό το επίδομα αναπηρίας που δεν έφυγαν όμως ποτέ από τη Δανία και αυτοί παίρνουν όλο το ποσό. Μετά υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία που επίσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 1408 κανονισμού και παίρνουν και εκείνοι το σωστό ποσό της σύνταξης αυτής. Η τρίτη ομάδα είναι Ευρωπαίοι πολίτες που διαμένουν νομοτύπως στη Δανία, που διέμεναν για πολλές φορές και για περίοδο 20 ετών στη Δανία, αλλά είναι από άλλα κράτη-μέλη. Εγώ είμαι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω και το δικό μου το παράδειγμα φωτίζει την κατάσταση. Οι δανεικές αρχές υπολόγισαν το ποσό στηριζόμενοι μόνο σε εσωτερικούς εθνικούς κανόνες. Και σύμφωνα με το 36.4 άρθρο πρέπει να ζητήσουμε ποσό ισοδύναμο με εκείνο που θα παίρναμε στην Πολωνία. Επίσης παραγνωρίστη ένα στοιχείο, το άρθρο 51 του κανονισμού 1408 ή το 50 4 ε, ε, του κανονισμού 883. Νομίζω ότι εν προκειμένου παραδιάστηκαν και οι δύο κανονισμοί. Επίσης αναφέρομαι στην ίση μεταχείριση και έλλειψη διακρίσεων. Έχουμε ένα παράδοξο εδώ. Άνθρωποι που δεν δούλεψαν ποτέ, άνθρωποι από τρίτες χώρες, νεότεροι μου κατά 20 χρόνια, οι οποίοι έλαβαν το επίδομα Παύλα Σύνταξη, η πλήρη. Όσοι προβλεπόταν την πήραν. Ενώ εγώ έζησα, εργάστηκα στη Δανία για 15 χρόνια και παίρνω πολύ μικρότερη σύνταξη. Άρα γίνονται διακρίσεις σε βάρος μου. Και είμαι και πιο ηλικιωμένη από τους άλλους. Δανείοι που δεν, υπήκοοι που δεν ε, δούλεψαν ποτέ παίρνουν 30.000, όχι 13 ενδεχομένως, ε, και εγώ παίρνω 8 και, κάποιες πρόσθε, και κάποια πρόσθετα επιδόματα που λαμβάνω από την Πολωνία, την πατρίδα μου. Όταν παίρνω δε το επικουρικό αν θέλετε από την Πολωνία, διαπιστώνω ότι τα εισοδήματά μου μειώνονται ακόμη περισσότερο και με το πρόσθετο αυτό ποσό. Α, θα χρειάζεται ένα συντονισμένο σύστημα. Η Γενική Αρχή δεν θα πρέπει να είναι να βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων και όχι να μειώνονται τα εισοδήματά τους. Επίσης θέλω να διαμαρτυρηθώ ενάντια στους κανόνες που ισχύουν για τον υπολογισμό των συντάξεων υπάρχει η δανεική παράγραφος 27α. Για δύο χρόνια ακούω ότι η κατάσταση δική μου δεν καλύπτεται από το άρθρο αυτό. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλαξε γνώμη και λέει ότι αυτό η πρόσθετη, αυτό το επικουρικό μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτού του κανονισμού και θεωρείται κοινωνικό, κοινωνικό βοήθημα πριν ε, να ε, αρχίσω να παίρνω ως ε, δικαιούμενα αυτή την σύνταξη αναπηρίας έπαιρνα μια, ένα άλλο επίδομα ανεργίας που επίσης ενέπιπτε στον 1408 και πριν από αυτό δούλευα με ευέλικτο ωράριο. Τα χρήματα που παίρνει κανείς από τα δύο αυτά επιδόματα μαζί ισούνται με την πλήρη σύνταξη επίδομα αναπηρίας που συνήθως ε, παίρνει ένας δανός υπήκοος. Η απάντηση λοιπόν που θέλω να πάρω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η εξής. Θέλω να ξέρω γιατί περίμενα 1,5 χρόνο στη Δανία για το συντονισμό των ε, συντάξεών μου. Δεν ε, σταθμίστηκαν, δεν ε, συντονίστηκαν μαζί με τα ποσά που παίρνω από την Πολωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου λέει ότι εμπίπτω στο πεδίο εφαρμογής ε, εθνικών κανόνων. Αυτό αντιβαίνει στους κανόνες, ούτε συνάδει με τα γεγονότα. Επίσης, η προϋπηρεσία, τα έτη προϋπηρεσίας, πώς υπολογίζονται. Και αυτό είναι άδικο. Εγώ θα πρέπει να πληρώ δύο προϋποθέσεις. Θα πρέπει να ζω τρία χρόνια τουλάχιστον στη Δανία πριν ζητήσω οτιδήποτε και η άλλη προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να δουλεύω ε, πλήρη απασχόληση επί 40 χρόνια. Ενώ οι Δανείοι πρέπει να πληρούν μόνο την δεύτερη προϋπόθεση. Μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι η, πρώτη προϋπόθεση βελτιώνει την κατάστασή μου. Ερωτώ όμως, γιατί δεν μπορώ να προσθέσω και άλλα 20 χρόνια που δούλεψα στην Πολωνία πριν μετακομίσω και εγκατασταθώ στη Δανία. Ε, δεν τους καταλαβαίνω αυτούς τους κανόνες. Νομίζω ότι είναι άδικοι. Δεν πρέπει εγώ να παίρνω λιγότερα χρήματα για όλα τα ε, χρόνια που εργάστηκα και πλήρωσα τους φόρους μου πάντοτε, ε, τις εισφορές μου και δεν με νοιάζει αν θα είναι επικουρικό ή πώς θα το πείτε ή αν θα συντονιστεί μαζί με την άλλη σύνταξη ή αν θα προσθεθούν όλα τα έτη προϋπηρεσίας μου. Δεν με νοιάζει, αλλά εκείνο που σας λέω είναι ότι εγώ μόλις τα βγάζω πέρα. Είμαι στο όριο της φτώχειας. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στη ε, Δανία όπως εγώ και υφίστανται τις ίδιες διακρίσεις που υφίσταμαι και εγώ. Επίσης υπάρχει και ένα παράρτημα ε, όπου οι δανεικές αρχές καταχωρούν έναν μεγάλο αριθμό ε, νομικών πράξεων που ισχύουν στην περίπτωσή μου και θα δείτε εκεί στο παράρτημα αυτό και μια, ένα νόμο δανεικό όπου αναφέρουν το ποσό της σύνταξης και υπάρχει ένα ποσό μόνο που αναγράφεται εκεί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι η ελάχιστη σύνταξη που δικαιούται κάποιος που παίρνει αυτή τη σύνταξη ε, αναπηρίας. Και επίσης έχουμε και το άρθρο 27α, όπου διαβάζουμε ότι το άρθρο αυτό θα εφαρμόζεται σε ανθρώπους όπως εγώ. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί επί χρόνια μου έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν εφαρμόζεται, δεν είναι στην περίπτωσή μου και μετά άλλαξε γνώμη. Και ακούω ότι μπορεί αυτό να είναι το ελάχιστο επίπεδο εσόδων όλων όσου διαμένουν στη Γαλλία που είναι 10.000 δανεικέ κορώνες. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν, εγώ έζησα 15 χρόνια στη Δανία, δούλεψα 20 χρόνια και γιατί δεν πληρώνομαι με το, την ίδια σύνταξη όπως άλλοι, το ίδιο ποσό. Δηλαδή, τι συντονισμός είναι αυτός μεταξύ Πολωνίας και Δανίας. Πρέπει να απογορευτεί αυτός ο συντονισμός, γιατί χωρίς το συντονισμό θα παίρνω περισσότερα η Κομισιόν Ο κύριος Φίλιξ Σάτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την αναφέρουσα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε εδώ ότι οι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων είναι πάρα πολύ περιορισμένε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απλώ αρμόδια για τον συντονισμό και όχι για την εναρμόνιση ε, συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Στην περίπτωση λοιπόν της αναφέρουσας, το επίπεδο των ε, παροχών εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από τα κράτη-μέλη. Το κοινοτικό δίκαιο δεν προβλέπει κανένα απολύτως επίπεδο παροχών. Το δικαστήριο στην πάγια νομολογία του επιβεβαίωσε ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Ο συντονισμός είναι το μόνο που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η μόνη της αρμοδιότητα. Δεν έχει αρμοδιότητα εναρμόνισης. Η μόνη απόφαση που ενδεχομένως μπορούμε να αναφέρουμε εδώ είναι η απόφαση του δικαστηρίου όπου αναφέρει το κοινοτικό δίκαιο δεν προσφέρει καμία εγγύηση όσον αφορά τη δραστηριότητα από το ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο που ενδεχομένως μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις ε, στα εισοδήματά τους και όχι αρνητικές. Δεν είναι δηλαδή ουδέτερη η μεταφορά δραστηριότητας από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Οι δύο αναφέροντες ε, αναφέρουν ότι δεν έχουν λάβει το πλήρες επίδομα αναπηρίας βάσει του νόμου της Δανίας. 49.08 του 71. Ο κανονισμός αυτός προβλέπει ότι ένας εργαζόμενος έχει δικαίωμα για επίδομα σύνταξης είτε ε, επίδομα αναπηρίας βάσει των ετών που εργάστηκε στη χώρα. Στην περίπτωση της αναφέρουσας υπάρχει ο χρόνος που εργάστηκε στην Πολωνία και ο χρόνος που εργάστηκε στην Δανία, βάσει των οποίων πρέπει να υπολογιστεί το επίδομα αναπηρίας. Βάσει ε, αυτή, αυτού του υπολογισμού ακριβώς το ίδιο πρέπει να ισχύει και για το επίδομα στην Πολωνία και για το επίδομα στη Δανία που σημαίνει βεβαίως ότι θα μπορούσε να ζητήσει δύο πλήρη επιδόματα αναπηρίας ή να ε, έχει το επίδομα αναπηρίας όταν ζει στην Δανία από τις δανικές αρχές και το αντίστοιχο όταν ζει στην Πολωνία. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα παροχών στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να δούμε το επίπεδο σε σχέση με το ε, βιωτικό επίπεδο της χώρας στην οποία διαμένει ο Ευρωπαίος πολίτης. Αυτό βεβαίως όμως είναι κάτι που δεν αφορά το κοινοτικό δίκαιο. Βάσει του άρθρου 26 για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης στη Δανία. Ήταν, ε, αν θέλετε, μια έρευνα που έγινε την πρώτη φορά που η αναφέρωσα ήρθε σε επαφή με τις υπηρεσίες της Επιτροπής και θεωρούμε ότι το επίδομα αυτό, η παροχή αυτή, μοιάζει με μία με ένα επίδομα, μία παροχή σε χρήμα. Και ότι ενδεχομένως μπορεί να υπολογιστεί και ένα συμπληρωματικό επίπεδο ε, επιδόματος, ένα συμπληρωματικό ποσό επιδόματος, το οποίο βεβαίως ενδεχομένως θα μπορέσει να το υπολογίσει το αρμόδιο κράτος μέλος και να το λάβει αναφέρουσα σαν επιπλέον ποσό. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να προσθέσουμε σαν συμπληρωματική παρατήρηση. Ευχαριστώ. Από ό,τι βλέπω δεν θα κάνει το άλλο στο λόγο. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον αναφέροντα. Έχετε το λόγο, το μικρόφωνο παρακαλώ και έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σα. Για να Ένα ερώτημα θα ήθελα να απευθύνω προ την Επιτροπή. Γιατί η πολωνική μου σύνταξη ε, δεν, ε, δεν υπάρχει συντονισμό μεταξύ της πολωνικής και της δανεική σύνταξη, μάλλον και γιατί δεν λαμβάνω τη συντάξη που λάμβανα ε, στο παρελθόν. Ε, δεν είπα ποτέ ότι θέλω να, ε, να λάβω δύο πλήρε συντάξεις και στην Πολωνία και στην Ενία. Βεβαίω και υπάρχει το άρθρο 50 του νέου κανονισμού και έχουμε και το άρθρο 51 που λέει ότι όταν λάβουμε σύνταξη από ένα κράτος μέλος θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός και επανυπολογισμό τη σύνταξη. Επανυπολογίζεται λοιπόν και καθορίζεται το νέο ποσό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της αναφερόμενη στη δεύτερη παράγραφο και ε, λέει ότι δεν δέχεται αυτό το άτομο παραπάνω χρήματα γιατί είναι δανή υπήκος. Αλλά εγώ θεωρώ ότι έχω τύχει ε, διακριτικής μεταχείρισης για τόσο καιρό που ε, απαιτώ μια ξεκάθαρη απάντηση. Βεβαίω και δεν μπορούμε να λάβουμε πλήρη σύνταξη και από τα δύο κράτη-μέλη, γιατί αν η Δανία αποδεχθεί τα χρόνια μου από την Πολωνία, τότε η Δανία μπορεί να, ε, αφαιρέσει το ποσό τη πολωνική σύνταξη. Ε, αυτό συμβαίνει συνήθω και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να συμβεί και στη δική μου περίπτωση. Ένα λεπτό έχετε εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Ευχαριστώ για το αν οι περίοδοι στην Πολωνία θα πρέπει να αναγνωριστούν από την Δανία, επαναλαμβάνω, όχι. Προφανώς η Επιτροπή δεν ε, λέει ότι η αναφέρουσα θέλει δύο ε, αλλά αυτό είναι το λογικό επακόλουθο αυτού του επιχειρήματος. Τώρα, γιατί δεν υπάρχει συντονισμό ανάμεσα στις δύο συντάξεις. Πρόκειται για... Ε, ε, ο όρος συντονισμό είναι ιδιαίτερα ευέλικτος. Τι σημαίνει στην πράξη. Σημαίνει ότι πρώτον μπορεί κάποιο να λάβει μια πολωνική σύνταξη στη Δανία. Ωστόσο υπάρχει ένας αρμόδιος κανονισμός που ε, προβλέπει έναν υπολογισμό, νέο υπολογισμό και έτσι Ελαμβάνεται υπόψη το γεγονό ότι αναφέρουσα ε, λαμβάνει σύνταξη σε άλλη χώρα. Ωστόσο, ο κανονισμό αναφέρει συγκεκριμένα ότι στι περιπτώσει όπου μόνο το εθνικό ε, επίδομα είναι ε, ανώτερο από αυτό το επαναπροσαρμοσμένο, αν θέλετε, επίδομα, τότε υπάρχει ο Η προσαρμογή λοιπόν του, προ... του επιδόματος δεν θα ήταν προς όφελός της. Θα ήταν σε βάρος της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ακούστηκαν όλα τα επιχειρήματα. Δεν μπορώ να σας δώσω ξανά τον λόγο. Τα έχουμε συζητήσει αυτά τα ζητήματα και στο παρελθόν, σε άλλες αναφορές. Ε, αυτό το ζήτημα αποτελεί απολυπιστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και των υπηρεσιών. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ε, κινούνται χωρίς ε, να χάνουν τα δικαιώματά τους. Αυτό πάντα στην Ευρώπη των 27. Από, τη, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατανοώ ότι δεν υπάρχουν πολλά μπορούμε να κάνουμε. Δυστυχώ θα πρέπει να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Προτείνω όμω στου συναδέλφου μου, αν και συμφωνείτε μαζί μου, να εξετάσουμε όλες τις προηγούμενες αναφορές για αυτό το ζήτημα και να επισημάνουμε αυτά τα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξανά. Να περιγράψουμε λοιπόν τα υπάρχοντα προβλήματα και ίσως μπορούμε ε, να επιστήσουμε την προσοχή των 27 κρατών μελών σε αυτά τα ζητήματα για να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό βέβαια, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη. Ευχαριστώ την αναφέρουσα. Προχωρούμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής σας διάταξης. Δύο αναφορές ε, έχουμε υπό το σημείο 29 του Μη Καλεράκη και τη Ιρένα Ρογκόφσκα Πολωνική Ιθαγένεια εξ ονόματο τη ε, Ένωση για την Πάυση τη Υπαίθρια Εξόριξη σε υπαίθριο λιγνητορυχείο στην νότια Συλλησία της Πολωνίας. Η κυρία Ρογκόφσκα είναι εδώ, έχετε το λόγο. Λέγω Μιρένα Ρογκόφσκα και υπέβαλα την υπαρίθμου 46-2010 αναφορά και εκπροσωπώ τους κατοίκους της περιοχής ως επικεφαλής στην ε, ε, πιτροπή για να σταματήσει το ρηχείο. Ε, υπάρχουν και εκπρόσωποι της περιφέρειας, εκπρόσωποι της Greenpeace. Στις 25 Ιανουαρίου μπόρεσα να υποβάλω την υπόθεση στην Επιτροπή, να την παρουσιάσω και υπενθυμίζω ότι η αναφορά αφορά την μη τήρηση των αποτελεσμάτων των δημοψηφισμάτων από 27 Σεπτεμβρίου 2009. Αυτό ήταν το δημοψήφισμα που αφορούσε τα σχέδια για τη δημιουργία ανοιχτού λιγνητορυχείου στην περιοχή που είναι στην κάτω Σιλεσία. Θέλω να ενημερώσω στην Επιτροπή ότι κανένα από τα αιτήματά μας δεν έγινε σεβαστό εντωμεταξύ και οι λόγοι για την υποβολή της αναφοράς εξακολουθούν να υφίστανται. Η κατασκευή του μεγάλου λιγνητορυχείου ανοιχτό εξακολουθεί να μας απειλεί και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί γιατί οι δραστηριότητες της πολωνικής κυβέρνησης σε συνοπτική νομοθετική διαδικασία σημαίνει ότι είμαστε στο παραπέντε να ε, προστατευτούν τα κοιτάσματα για, και αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσει η εξόρυξη. Αυτό ε, ανεξάρτητα από το αν θα κατασκευαστεί το συγκεκριμένο λιγνητορυχείο ή όχι. Και αυτό αντιβαίνει στις ε, αποφάσεις των τοπικών αρχών ε, και των δημοτών που ψήφισαν στο δημοψήφισμα. Η χώρα μας έχει λόγο να περηφανεύεται όταν πρόκειται για κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές. Προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά που τη χωρίζουν από την Δύση. Αλήθεια είναι όλα αυτά. Να θυμόμαστε όμως ότι προκειμένου περί εξόρυξης άνθρακα ελιγνίτη. δεν θέλει η χώρα μας να προχωρήσει ε, και να χρησιμοποιήσει προηγμένες τεχνολογίες και παραβιάζει κανόνες, παρακάμπτει το δίκαιο. Οι πολίτες λοιπόν ρωτούν γιατί μας αγνοείται, γιατί δεν μας μιλάει κανείς, γιατί δεν θέλει κανείς να απαντήσει στα αιτήματά μας εμείς ε, ε, δεν θέλαμε να συζητήσουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα στις Βρυξέλλες. Ελπίζαμε δε ότι μετά την ε, παρέμβασή μας ε, τον Ιανουάριο θα μπορούσαμε εσωτερικά να λύσουμε το πρόβλημα. Καλέσαμε και τον Πολωνό Πρωθυπουργό να επισκεφθεί την περιοχή μας. Αλλά ο Πρωθυπουργό μας αγνόησε και δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο... Δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βρει και χρόνο να μας ε, ακούσει, ενώ μας άκουσε, ενώ ο Πρωθυπουργό όχι, ή ο Οι πολωνικές αρχές θέλουν να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των εταιριών σε βάρος χιλιάδων πολιτών που ζουν εκεί, σε βάρος του περιβάλλοντος εκεί. Ε, έγιναν και άλλα παρόμοια δημοψηφίσματα σε άλλες περιοχές της γενικότερης περιφέρειας της κάτω Σιλεσίας και παρά τις υποσχέσεις ότι θα ε, γινόντουσαν σεβαστά τα αποτελέσματα, δεν έγιναν. Υπάρχει δε μία διάταξη που προβλέπει ότι οι αρχές πρέπει να προστατεύουν τα κοιτάσματα λιγνίτη. Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος το Μάρτιο ενημέρωσαν τις ειδικές μας τοπικές αρχές σχετικά με την αποδοχή του γεωλογικής τεκμηρίωσης για τα κοιτάσματα λιγνίτη και υπάρχει η απειλή που όλο και μεγαλώνει τώρα. Γι' αυτό αρχίσαμε την εκστρατεία και είπαμε ανάπτυξη ναι, ανοιχτό ορυχείο λιγνίτη όχι. Αυτή η εκστρατεία εκπροσωπείται από την περιφέρεια που κατοικείται από 100.000 ανθρώπου και οικολογικέ οργανώσεις, πράσινε οργανώσει, οι οργανώσει των πολιτών. Όλοι συμμετέχουν σε αυτή την εκστρατεία. Είναι μαζική ε, από κάτω προ τα πάνω κίνηση αυτή των πολιτών και είναι και η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Εμείς κάνουμε εκστρατεία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλουμε οικονομίες χαμηλής ε, χαμη, ε, κατανάλωσης άνθρακα ε, χαμηλών εκπομπών ρήπων. Αυτά είναι τα επιχειρήματα. Άλλα δεν έχουμε για να δώσουμε στις αρχές. Και η βοήθειά σας, η βοήθεια κάθε ευρωβουλευτή είναι πολύτιμη. Έχουμε τόσους πολλούς που διαμαρτύρονται και είμαστε και πολλοί. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η υπόθεσή μας είναι εξαιρετική γιατί πρόκειται για ε, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ε, συμβολίζουν το μέλλον. Είναι το μέλλον. Θέλουμε λοιπόν η Επιτροπή Αναφορών να το εξετάσει το θέμα, να κάνει μια διαρευνητική αποστολή και μια κοινοβουλευτική έκθεση που θα περιέχει προτάσεις και ελπίζομαι ότι θα ψηφιστούν και από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να πιέσουμε τις τοπικές αρχές να αρχίσουν διάλογο με τους πολίτες τους ε, και πριν από την ε, Προεδρία από την Πολωνία της Ένωσης. Ευχαριστώ. Και τώρα η Κομισιόν, ο κύριος Μπρίκλαντ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η υπόθεση αυτή αφορά ένα στρατηγικό σχέδιο στην Πολωνία που ουσιαστικά παγώνει κάποια αποθέματα άνθρακα σε ορισμένες περιοχές πάγωμα όσον αφορά τη χρήση αυτών των κοιτασμάτων λιγνίτη και προηγουμένως έγινε μία βεβαίως στρατηγική μελέτη αντικτύπων Θελήσαμε λοιπόν να δούμε καταρχήν την συμβατότητα με τις κοινωτικές οδηγίες. Δεν βρήκαμε παραβιάσεις όσον αφορά τη διαδικασία που έχει αποφασιστεί και η βασική <clears throat> διαμαρτυρία των αναφερόντων είναι ότι δεν είχαμε χρόνο να σχολιάσουμε. Εμείς ε, σχολιάσαμε και δεν νομίζω ότι μπορείτε να πείτε ότι δεν υπήρξε διαβούλευση από τη στιγμή που οι τοπικές αρχές γνωρίζουν πολύ καλά τη θέση τη δική σας. Μέχρι το 2013 δεν θα γίνει τίποτα. Η ενημέρωση έχει ξεκινήσει και θα πρέπει εδώ να σας πω ότι δεν έχουμε εντοπίσει παραβίαση. Προς το παρόν τουλάχιστον. Εάν κάτι αλλάξει, εάν ε, γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που μας ανέφεραν οι πολωνικές αρχές, φυσικά και θα ξαναρχίσουμε την έρευνα. Προς το παρόν παγώνει η χρήση των ε, κοιτασμάτων λιγνίτης, δεν υπάρχουν προβλήματα με το περιβάλλον. Τουλάχιστον η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος διαπίστωσε ότι αν κάποιος παγώσει δραστηριότητες μέχρι το 2013 μπορεί να υπάρξουν όντως κάποιες αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την ιδιοκτησία στην περιοχή. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό που μπορέσαμε να διαπιστώσουμε. Αλλά κατά τα άλλα δεν είδαμε όπως σας είπα παραβίαση της οποιασδήποτε οδηγίας. Οι αρχές της Πολωνίας σας έχουν απαντήσει και η Επιτροπή πιστεύω θα πρέπει να συνεχίσει να παίξει ενεργό ρόλο στην υπόθεση αυτή. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη από την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στηρίχθηκε σε ευσεβείς πόθους τροποντινά. Όταν βλέπω τα πολωνικά έγγραφα, βλέπω ότι λέει ότι διεξήχθη ε, κοινωνικός διάλογος και κοινωνικές διαβουλεύσεις με ικανοποιητικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι το έργο έγινε δεκτό από τους κατοίκους της περιοχής. Όμως, στο δημοψήφισμα ξεκαθάρισαν οι κάτοικοι ότι δεν το θέλουν το ανοιχτό λιγνητο ρηχείο. Αυτό είναι παραπλανητικό. Και επίσης διαφωνώ με αυτά που είπε η Επιτροπή σχετικά με την ε, καταληκτική ημερομηνία του 2030, ενώ ή 13, δεν είναι σαφές αν ε, όμως παγώσουμε τα κοιτάσματα, αυτό σημαίνει ότι παγώνουμε την ανάπτυξη της περιοχής εν γέννη και αυτό σημαίνει ότι τα κονδύλια τα οποία εισέρευσαν στην υποδομή της περιφέρειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα χρήματα χάθηκαν σπαταλήθηκαν και λέει ότι θα είναι και το μεγαλύτερο ανοιχτό λιγνητορυχείο στην Ευρώπη. Και εμείς τώρα μιλάμε ε, και θεωρητικολογούμε για οικονομίες χαμηλού άνθρακα κλπ. Θα πρέπει, 2030, ε, πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεπείς ε, προς τις, στα υψηλά μας οράματα. 2030 είναι η καταληκτική. Τώρα, οι πολωνικές αρχές απάντησαν στην επιστολή και οι αναφέροντες δεν την έλαβαν. Η πολωνική κυβέρνηση απαντά λέγοντας ότι δεν υπονομεύει το δικαίωμα των ΟΤΑ να ε, κάνουν ε, σχέδια χωροταξίας. Αυτό είναι τελείως αντιφατικό, γιατί από τη μία πλευρά τα κοιτάσματα θα προστατευτούν και, από, και παγώνουν και από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση λέει όχι, οι τοπικές αρχές, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ε, απόλυτα ελεύθερα μπορούν να σχεδιάζουν την ανάπτυξη της περιοχή τους. Είναι σχιζοφρένη αυτό από την πλευρά της πολωνικής κυβέρνησης. Τι είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Και θα ήθελα να ρωτήσω και τη γνώμη της Greenpeace Επίσης πείτε μας εσείς τι πιστεύετε για το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ανοιχτό λιγνητορυχείο του κόσμου θα γίνει εκεί σε αυτή την περιοχή της Πολωνίας. Ευχαριστώ. Ε, εκπρόσωπος της ε, Δημοτικής Αρχής της Κουνίτσα. Ευχαριστώ που μου δίνατε το λόγο. Θα ήθελα να πω ότι βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, γιατί η Επιτροπή Αναφορών θα ήθελε να επιλύσει το ζήτημα αυτό, και η Επιτροπή είναι ένα μέσο ε, αν θέλετε, μεταξύ των διαφόρων μερών. Ο αναπληρωτής αντιπρόεδρος ε, της πολωνικής ε, κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι δεν θα κατασκευαστεί αυτό το ανοιχτό λιντορυχείο ε, σε εκείνη την περιοχή γιατί δεν υπάρχουν επενδυτέ. Επομένω, έχουμε αυτή την πληροφόρηση και ξέρουμε ότι δεν θα κατασκευαστεί αυτό το λιντορυχείο. Και αυτό είναι κρίσιμη σημασία. Κάτι άλλο που είναι κρίσιμη σημασία είναι ε, η πράσπιση των συμφερόντων ε, των πολιτών, χιλιάδων πολιτών που βρίσκονται εκεί, σε αυτή την περιοχή. Και βεβαίως και υπάρχει έλλειψη διατάξεων που ε, προσπίζονται την διατήρηση των, των κοιτασμάτων. Γιατί Τίποτα δεν μπορεί να γίνει, ε, δεν μπορούν να κατασκευαστούν σχολεία, νοσοκομεία, κατοικίες και το καθεξής, εφόσον η πολιτική κυβέρνηση εμένει σε, σε αυτές τις αρχές και αυτές τις διατάξεις. Ε, υπάρχει ένα σχέδιο κατασκευής ενός ε, δρόμου στην περιοχή, αλλά και αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα μα έχει πει η πολιτική κυβέρνηση που μιλάει για προστασία των ε, κοιτασμάτων. Από την άλλη όμως θέλουν να, να κατασκευάσουν αυτοκινητόδρομο εκεί πέρα. Σε όσα μας είπε η θα ήθελα να, να, μάλλον, να απευθυνθώ στην Επιτροπή και να την καλέσω να ζητήσει γραπτή επιβεβαίωση από τον εκπρόσωπο τη πολιτική κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να κατασκευαστεί το γνητορυχείο σε εκείνη την περιοχή. Ότι δηλαδή αυτό που ο κύριο Παύλακ είναι αλήθεια. Να καλέσουμε επίση την πολιτική κυβέρνηση να μα πει εάν θα ε, συνεχίσει αυτή η διατήρηση των κοιτασμάτων ή όχι. Έχουμε βέβαια λάβει πληροφορίες, αλλά όχι γραπτός. Εάν ε, λάβουμε θετική, θετική απάντηση, δεν υπάρχει προστασία κοιτασμάτων, δεν υπάρχει ορυχείο. Και έτσι λύνεται το ζήτημα διαπαντός. Η Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να ζητήσει άμεσα ε, την ε, πολωνική κυβέρνηση γιατί οι πολωνικοί αξιωματούχοι τα έχουν πει αυτά αλλά θα πρέπει να μας τα επιβεβαιώσουν και γραπτός. Αυτή είναι η πρότασή μου προς την Επιτροπή. Η Κομισιόν θα πρέπει να έρθει σε επαφή ε, με τις ε, πολωνικέ αρχέ και έτσι μπορεί να επιληθεί μια για πάντα αυτό το ζήτημα. Μια ερώτηση. Ποιο είναι, ποιος είναι ο ρόλο τη Greenpeace σε αυτή την υπόθεση. Γιατί βλέπω για την πρώτη φορά συμμετέχει η Greenpeace σε τέτοιο ζήτημα. Ευχαριστώ, συνάδελφο Ποσνάρο. Ευχαριστώ. Είναι λίγο συγκεχημένη η κατάσταση. Με μία ανεπίσημη, αν θέλετε, δήλωση του αναπληρωτή Πρωθυπουργού για το σχέδιο αυτό και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι ο πιο επίσημος ε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ εν ώψη της Επιτροπής Αναφορών που μας λένε ότι οι πολωνικές αρχές τους έχουν ενημερώσει ότι δεν θα ξεκινήσει τίποτα, ότι δεν έχει ξεκινήσει τίποτα και μέχρι το 2013 δεν θα γίνει τίποτα και αν ποτέ ξεκινήσει κάποιο σχέδιο θα διασαφινιστεί προηγουμένως η υπόθεση. Γιατί να μην προβλέψουμε αλλά να αντιδράσουμε εκ των υστέρων. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλον προσπαθεί να διορθώσει κάποια πράγματα ενώ είναι πολύ αργά. Μήπως θα ήταν καλύτερα να έχετε μία προληπτική δράση καταρχήν ζητώντας πληροφορίες από τα κράτη-μέλη πριν ξεκινήσει ένα τέτοιο σχέδιο. Εδώ σαφώς και χρειάζεται μια στρατηγική μελέτη αντικτύπου, αξιολόγηση αντικτύπου. Οι πληροφορίες σας είναι ελάχιστες. Δεύτερον, τι νόημα έχει να υπάρχει δημόσια συζήτηση και διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ αγνοούνται τα δημοψηφίσματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούμε τους πολίτες της περιοχής να λένε ότι δεν θέλουν την ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών που θεωρούν ότι έγινε δημόσια διαβούλευση και ο κόσμος είναι πανευτυχής. Εγώ ακούω την πρόταση του κυρίου του συναδέλφου, που ζητά αποσαφήνιση της κατάστασης το συντομότερο δυνατών και τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσει μια αξιόπιστη επίσημη απάντηση και να κλείσει η αναφορά εάν ε, πρέπει να κλείσει και να ικανοποιήσουμε τους αναφέροντες οι οποίοι ήρθαν εδώ γεμάτοι προσδοκίες και ελπίδες. Σας ζητώ λοιπόν κυρία Πρόεδρε να στείλετε το αίτημά μας εξ ονόματος Επιτροπής Αναφόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κυβέρνηση της Πολωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Στηρίζω απολύτως αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Um, θα δώσω ε, ένα λεπτό να απαντήσει η αναφέρουσα και μετά θα πρέπει να κλείσουμε, να τελειώσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνούμε με την πρότασή σας. Θα ήταν αυτό μία λύση στο πρόβλημά μας. Επίσης ρωτάτε γιατί συμπεριελήφθη στη διαδικασία η Greenpeace. Ίσως αυτό το λεπτό μπορούμε να το δώσουμε στον εκπρόσωπο της συγκεκριμένης οργάνωσης. Ο κύριε Γιάρ, θα φύγουν ε, οι διερμηνείς 30 δευτερόλεπτα. Συμφωνείτε με την πρόταση. Α, ας ολοκληρώσουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Δεχόμαστε την πρόταση όλοι. Θα ζητήσουμε διευκρινήσεις επί όλων των θεμάτων από τις πολωνικές αρχές, όλα σε όσα αναφέρθηκε και αναφέρουσα και θα επανέλθουμε όταν απαντήσουν οι πολωνικές αρχές. Ευχαριστώ και λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς για το πρόσθετο χρόνο που μας έδωσαν. 25, 27, 40, 42, 51 και 60 αναφορές θα παραμείνουν ανοιχτές. Ευχαριστώ.